Καλησπέρα σας. Παρακαλώ θερμά τους προσκεκλημένους μας να καθίσουν γιατί θα θέλαμε να αρχίσουμε την δημόσια κρόασή μας. Let the... Σας καλωσορίζω λοιπόν στη δημόσια κρόαση με θέμα την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι μια ακρόαση που οργανώνει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων. Όπω θα γνωρίζετε, στο ψήφισμα του, 2010 για την κατάσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ένα νέο πλαίσιο, να χρησιμοποιήσουν μάλλον το νέο πλαίσιο της συνθήκης Λισαβόνας για να εφαρμόσουν μια περιεκτική πολιτική ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα εξασφαλίζει ε, μηχανισμούς αποτελεσματικούς για να αποτραπούν ή να αντιμετωπιστούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, γιατί έχω την τιμή να προεδρεύω τη σημερινή, τη σημερινή συνεδρίαση γιατί ήμουν και εγώ εισηγήτρια, συνεισηγήτρια στο σχετικό ψήφισμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να παρακολουθούμε την κατάσταση για τα θεμελιώδη δικαιώματα χρόνο με το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της δημόσια αυτής ακρόαση για την εφαρμογή του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι να αξιολογήσουμε τις τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αφορά την προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Προσβλέπω σε μια καρποφόρα συζήτηση και καλωσορίζω θερμά εδώ και ε, ευρωπαϊκούς φορείς, διεθνούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκπροσώπους ε, ε, οργανώσεων και ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε ένα υπερφορτωμένο πρόγραμμα και πολύ ενδιαφέροντες προσκεκλημένους. Έχουμε υψηλέ προσδοκίες λοιπόν και για την ποιότητα των ομιλιών και των παρεμβάσεων σας θέλω παρακαλώ όλους να τηρήσετε ευλαβικά το χρόνο σας, το χρόνο αγόρευσης, για να προλάβουμε και να τελειώσουμε εγκαίρος στις 6.30. Στόχο είναι η προώθηση, επαναλαμβάνει και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο τμήμα τη ε, δημόσια Το δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με την ένδικη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο τρίτο μέρος το πρόγραμμα δράσης πολιτών για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μετά από κάθε τμήμα της δημόσιας ακρόσης θα γίνει συζήτηση. Γι' αυτό και θα ήθελα παρακαλώ όσοι λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση να παρουσιάζουν τον αυτό τους και να σημειώνουν αν θέλουν να λάβουν το λόγο και αναφέροντας και το όργανο που εκπροσωπούν στο κατάλογο που θα κυκλοφορήσει για να συμπληρώσουμε το κατάλογο με τους ομιλητές. Θα ήθελα να δώσω το πρώτο το λόγο στην κυρία Μόνικα Φλασίκοβα Μπένοβα, που είναι η συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση προστασία θεμελιώδων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μα κάνει την εισαγωγική παρουσίαση. Κυρία Μπένοβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ και του συμμετέχοντε, κυρίε και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει όλο και μεγαλύτερη σημασία στα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν είμαι υπέρ των υπερβολών και των βαρύγδουπων ε, εκφράσεων, αλλά μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής η ιδέα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Ένωσης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Γι' αυτό και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που ανέλαβα την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισθάνομαι και ιδιαίτερη χαρά για τη συμμετοχή μου στη σημερινή αυτή δημόσια ακρόαση. Όπως ξέρετε όλοι, η διεξαγωγή της δημόσιας ακρόασης ήταν και ο λόγος αναβολής της έκθεσης για το 2012, γιατί περιμένουμε τις παρατηρήσεις από την ακρόαση αυτή και τις διάφορες παρεμβάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την εκπόνηση της έκθεσης, γιατί τα μέχρι στιγμής έγγραφα που είχαμε δεν ήταν επαρκή. Και ούτε η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε το, η μελέτη που είχε περιεκτικές πληροφορίες για την κατάσταση των δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη και τον αντίκτυπο της ε, συνθήκης στο χάρτη ήταν επαρκή στοιχεία. Θα εξετάσουμε και τα θεσμικά και τα διαδικαστικά ζητήματα γιατί έχουν, έχει τροποποιηθεί το πλαίσιο γι' αυτό και τώρα θα δώσουμε έμφαση στα πιο ουσιαστικά σημεία. Η ετήσια έκθεση λοιπόν θα πρέπει να περιλαμβάνει και νέα στοιχεία προκειμένου να τροφοδοτήσει τη συζήτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και να μην αποτελεί μια στήρε επανάληψη των προηγούμενων εκθέσεων. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για σχετική νομολογία αλλά και για έμπρακτες πτυχές της εφαρμοσιμότητας των ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο έργο προϋποθέτει στενές επαφές και με τους ε, διαφορούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Έτσι θα συγκεντρώσουμε εγκαίρως ε, χρήσιμες πληροφορίες. Αλλιώς ε, θα είναι μια έκθεση που απλώς θα διαπιστώνουμε την τρέχουσα κατάσταση στα θεμελιώδη δικαιώματα και θα υπογραμμίζουμε τα ακολουθητέα βήματα. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Έχουμε υψηλότερε φιλοδοξίες. Κάθε η έκθεση πιστεύω ότι θα πρέπει να αξιολογεί την πρόοδο από την ανάληψη των δεσμεύσεων στην εφαρμογή και να δίνει μια απάντηση στον προβληματισμό των ενδιαφερομένων. Μόνο έτσι θα ανακτήσουμε και τις, την ελεγκτική μας αρμοδιότητα και την αρμοδιότητα της αξιολόγηση από το να παρουσιάζουμε ένα απλό ευχολόγιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ όχι μόνο τους εκπροσώπους των κοινωτικών θεσμικών οργάνων, αλλά και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως είναι η Κοινωνική Πλατφόρμα ή η η διεθνη Αμνηστία, το Ευρωπαϊκό Γραφείο, μεταξύ άλλων. Οι ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκπροσωπούν πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει επαρκή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προσβλέπουν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλώντας το να αντιδράσει στις ε, πολιτικές διακηρύξεις και πρωτοβουλίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χρειάζονται συζητήσεις ε, γιατί θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις για το τι θα πρέπει να αλλάξει και ποια είναι η ακολουθητέα οδός. Η δημόσια αυτή ακρόαση και η ετήσια έκθεση που έχω την τιμή να προετοιμάσω θα αποτελέσουν την ευκαιρία για τη συζήτηση αυτή στην οποία θα συμμετέχουν ενεργά και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Επίσης δίνεται εξέχον ρόλος τι ε, εθνικέ οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα εθνικά θεσμικά όργανα που δίνουν σωστέ πληροφορίε για την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Παρόλο που μέχρι στιγμή δεν είχαν ποτέ αναμειχθεί σε δημόσιε ακροάσεις τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Χαίρομαι λοιπόν γιατί σήμερα έχουμε και εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τις Εθνικές Οργανώσεις μάλλον, τις Εθνικές Οργανώσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. και μας ενδιαφέρει και η δική τους ε, γνώμη. Θα πρέπει να εξετάσουμε τη διαδικασία, μια διαδικασία που θα είναι παρόμοια με αυτή με την ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή ε, ζητώντας από την Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της. Μπορούμε να ζητούμε και πιο τακτική αξιολόγηση από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά και μπορούμε να ζητούμε και γνωμοδοτήσει ε, των νομικών υπηρεσιών για το πόσο είναι συμβατέ οι εθνικέ νομοθεσίε με το χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα μπορούμε επίση να διοργανώνουμε και ετησίω ε, διασκέψει στη συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσει και διεθνεί φορεί πέραν της δημόσια ακρόση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τις διαδικασίες επί παραβάση και να εξασφαλίσει έμπρακτη προστασία και προώθηση των θεμελιδών δικαιωμάτων και να έχει πιο συστηματική διαβούλευση με τη, τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να συμμετέχει πιο ενεργά σε διάλογο με το Κοινοβούλιο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσει και σημαντικό οργανισμό που θα έχει συντονιστικό ρόλο μεταξύ των αντίστοιχων θεσμών των, κρατών μελών. Θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση και τέλος να επικεντρωθούμε και στο, στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Χρειάζεται συζήτηση για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ενεργούς δέσμευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, και διαβουλεύσεις με κοινωνία των πολιτών και με κυβερνητικές ε, οργανώσεις σε προκατακτικέ φάσει νομοθετική διαδικασία, αλλά και στην εκπόνηση μελέτη επιπτώσεων ε, των νομοθετημάτων σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Διαβάζοντα το πρόγραμμα τη δημόσια ακρόαση και του κορυφαίου προσκεκλημένου μα, Είμαι βέβαιη ότι η δημόσια αυτή ακρόαση θα παίξει κρίσιμο ρόλο και θα βοηθήσει στην επιτυχία της ετήσιας έκθεσης. Περιμένω λοιπόν τα αποτελέσματά της. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπένοβα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Πολ Νέμιτς, που είναι διευθυντής για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ηθαγένεια. Έχετε το λόγο κύριε Νέμιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να διαβεβαιώσω την εισηγήτρια, την κυρία Μπένοβα, πως βεβαίως αναμένουμε τη συνεργασία μαζί της και νομίζω πως μπορώ να πω πως ε, το να δοθεί η ζωή στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το να μπορέσουν οι πολίτες μας να εκμεταλλευτούν τα δικαιώματα ε, που περιγράφει ο χάρτης νομίζω είναι βασικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την πρόοδο που έχει σημειωθεί από όταν κατέστη δεσμευτικός ο χάρτης. Πρώτα απ' όλα, τακτοποιήσαμε τα του οίκου μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του χάρτη και έχουμε αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές ε, για τους υπαλλήλους μας που ε, νομοθετούν, ε, εμπλέκονται στην νομοθετική διαδικασία Καλό είναι πάντα να ξεκινάει κανεί από τα του οίκου του. Δεύτερον, το Συμβούλιο δεσμεύτηκε το Φεβρουάριο του 2011 να καταβάλει αυξημένε προσπάθειες να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως περιγράφονται στο χάρτη. Και θα ήθελα να σα δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Τι διαφορά έχει ήδη κάνει ο χάρτης αυτός όσον αφορά τι νομοθετικές προτάσεις και τι επίτευγμα είναι και μην ξεχνάμε βεβαίως την γέννηση αυτού του χάρτη, την εμπλοκή των βουλευτών και των κρατών μελών, τη συνέλευση, ένα μεγάλο επίτευγμα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ένα παράδειγμα λοιπόν των μορφή προτάσεων της Κομισιόν. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στη διαφορά μεταξύ μια πρότασης του 2008 για να επιτραπεί στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν σαρωτέ σώματος και μετά την πρόταση του 2011. Στην τρέχουσα πρόταση έχουμε ε, την προστασία της χάρτης, οπότε απαγορεύονται ρητά οι χάρτες με ακτίνες και θα έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν το να υποστούν αυτή τη σάρωση οι επιβάτες. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν θα υπήρχαν χωρίς το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και είναι βεβαίως επίτευγμα του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας, κάτι το οποίο δείχνει πρακτικά αποτελέσματα του χάρτη ε, επί της νομοθεσίας. Τώρα, όταν μιλάμε για τα δικαιώματα και τον πρακτικό αντίκτυπό του στη ζωή των πολιτών. Πρέπει να δούμε το τι κάνουν τα δικαστήρια. Γιατί βεβαίω τα ατομικά δικαιώματα πάντα θα πραγματοποιούνται μέσω των δικαστηρίων. Ούτε η Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο θα κάνει κάτι. Μάλιστα μέσω της ε, διαδικασίας επί παραβάση, η Κομισιόν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και η απόφαση του Εθνικού Δικαστηρίου δεν ε, αποδίδει δικαιώματα σε ένα άτομο. Αυτό γίνεται μέσω της απόφασης του Εθνικού Δικαστηρίου. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μοιράσετε αυτό το, να, το μήνυμα, να ενημερώσετε τους εθνικούς δικαστές, ε, τους ε, δικηγόρους ε, στις χώρες σας ε, όσον αφορά την ε, νομολογία και την ισχύ του ευρωπαϊκού δικαίου. Και βλέπουμε ήδη κάποιο βαθμό διείσδυσης που είναι μια αρχή και νομίζω μπορεί να δημιουργήσει ελπίδες πως τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Το 2009 μόνο δύο αιτήματα είχαμε από εθνικά δικαστήρια μία πρώτη ε, προκαταρκτική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από αίτημα ε, του, των Εθνικών Δικαστηρίων αριθμοί οι οποίοι αυξάνονταν ήδη το πρώτο εξάμεινο του 2011 είχαμε 20 τέτοια αιτήματα από εθνικούς δικαστές για ε, προδικαστικά ερωτήματα. Οπότε, έχουμε αρκετά μεγάλη πρόοδο και νομίζω μπορούμε να δικαιολογήσουμε μια πορεία. Και έχουμε ήδη και αποφάσεις πέρα από τα προδικαστικά ερωτήματα. Θα αναφέρω την απόφαση σε Γιάιφερτ και τεστ ΑΣΑ. Ταυτόχρονα νομίζω πως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όταν μιλάμε για το χάρτη, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα πολιτικής, δεν θα πρέπει να δημιουργούν βεβαίως ε, λανθασμένες προσδοκίες ε, στους πολίτες. Δεν θα πρέπει να λέμε υπερβολές, να λέμε πως η Ευρώπη θα λύσει προβλήματα εκεί που δεν έχει αρμοδιότητες. Γιατί έτσι τι θα γίνει, θα απευθυνθούν σε λάθος αρχές οι πολίτες. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ε, και ορθή, ειδικά όταν μιλάμε για πράγματα όπως το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και για το λόγο αυτό, η Κομισιόν ήταν σαφής στην ε, πρώτη έκθεσή της ε, του Μαρτίου του 2011 για την εφαρμογή του χάρτη και θα συνεχίσει να είναι σαφής γιατί βεβαίως ε, η υπευθυνότητα και η λογοδοσία σημαίνει πως δεν θα πρέπει να δημιουργούμε Λανθασμένε προσδοκίες. Είχαμε και ένα σεμινάριο με τους σα σας Επιτροπής Αναφορών πρόσφατα που εστίασε στα ατομικά δικαιώματα από τη δική μα Σκοπιά και στο πόρταλ ε, ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ε, θα δώσουμε πληροφορίες στους πολίτες που μπορούν να στραφούν στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τα ατομικά τους πια δικαιώματα. Οπότε μιλάμε για θεσμικά όργανα, ΜΚΟ και ε, κρατικούς φορείς πλην δικαστηρίων. Οπότε θα ήθελα να γίνει μια συζήτηση με όλους εσάς για το ποιο είναι η δυνατότητα αφενός των δικαστηρίων και αφετέρου συνήγορων του πολίτη κτλ. για να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Πρέπει να δούμε ολόκληρο το φάσμα θεσμικών οργάνων, να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά τους και να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει ο χάρτης αυτός για τους πολίτες μας. Τέλος, θα θέλαμε να Ε, παρουσιάσουμε και μια ετήσια έκθεση το 2012 και ελπίζω αυτό να αποτελέσει χρήσιμη βάση για τη δουλειά του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Νέμιτς, ο ε, επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τόμας Χάμαρμπεργκ, Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σας καλωσορίζουμε και πάλι και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στενά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με μία εξομολόγηση. Όταν γκούστηκε για πρώτη φορά η ιδέα ενός χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ευρωπαϊκή Ένωσης, εγώ ήμουν πολύ επιφυλακτικός, ήμουν κατά. Γιατί θεωρώ πως υπήρχε ήδη μία συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση και αν έπρεπε να γίνει κάτι άλλο θα έπρεπε να ε, σκεφτούμε πως είναι πολύ πιο οικονομική λύση να αναπτύξουμε την ΕΣΔΑ, ίσως άλλο ένα πρωτόκολλο. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος οι ίδιες χώρες να χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές συνθήκες. Βεβαίως όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης είναι και μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμμελούμενο μέρη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και βεβαίως δεσμεύονται να σέβονται τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φοβά, ε, φοβήθηκα πως θα δημιουργηθεί σύγχυση όσον αφορά τις αρμοδιότητες στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ε, μέρη είχα άδικο, αλλά νομίζω πως κάποια επιχειρήματα που είχα αναπτύξει τότε ισχύουν και νομίζω πως εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα έλλειψης συντονισμού μεταξύ των δύο αυτών δομών. Είχα τις προσωπικές μου εμπειρίες, οι οποίες ήταν κάπως απογοητευτικές. Παραδείγματος χάρη όταν συζητήσαμε τους νόμους ε, περί ΜΜΕ στην Ουγγαρία είδα πως ε, μπορούσαν νομίζω πιο αποτελεσματικά να κινηθούμε μέσω του Συμβουλίου της ε, Ευρώπης ενώ η Κομισιόν αντιθέτως μπήκε σε ένα διάλογο και μονοπόλησε το διάλογο, έτσι ήταν τουλάχιστον η άποψη στη Βουδαπέστη και έγιναν κάποιες λίγες αλλαγές, όχι πολύ θεμελιώδεις, από το Κοινοβούλιο και η ατμόσφαιρα ήταν ότι εντάξει τώρα τα προβλήματα λύθηκαν όσον αφορά τις αντιδράσεις στην Ευρώπη. Είχαμε όμως ουσιαστικές αντιρρήσεις ε, όσον αφορά και άλλες αλλαγές του νόμου, οπότε εκεί πέρα υπήρχε μια έλλειψη, θα έλεγα, συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων αυτών θεσμικών οργάνων. Σήμερα το πρωί γινόταν σε αυτό το κτίριο μια συζήτηση για τα προβλήματα όσον αφορά την προφυλάκηση και υπήρξε μια θαυμαστή πρωτοβουλία της κυρίας Ρέντινγκ ε, να αποστείλει μια πράσινη βίβλο για να ενθαρρύνει μια συζήτηση για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να μειωθεί ο κίνδυνος κατάχρησης του μέσου της ε, προφυλάκησης. Και έχουμε προβλήματα όχι μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ περισσότερο σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αλλά όταν ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως το ζήτημα αυτό δεν είναι καινούριο. Στην Ευρώπη υπάρχουν σαφείς διατάξεις για την προφυλάκηση στο άρθρο 5 της ε, ΕΣΔΑ που λέει πως εάν υπάρχει απόφαση περί προφυλάκησης θα πρέπει αυτή να επανεξετάζεται τακτικά και πως θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Και υπάρχει και νομολογία που νομίζω πως ε, ισχύει για όλα τα κρατη και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσταση από τους ε, υπουργούς που προσωπούν όλες τις κυβερνήσεις και τις άλλες ε, Ευρωπαϊκή Κοινωνία και των κρατών μελών και τι άλλε που αναφέρουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούν όταν αναλύουν το πρόβλημα τη ε, προφυλάξης. Και μετά υπάρχουν ε, διάφορε συστάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστήριων που επίση έχουν σημασία σε αυτή τη συζήτηση και πρέπει να γίνει ακόμα αρκετή δουλειά έτσι ώστε να φροντίσουμε πως όταν υπάρχει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα η εμπειρία που υπάρχει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ε, ΟΑΣΕ, δηλαδή και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, να διαμοιράζεται. Ε, θα πρέπει να το θεωρούμε αυτό ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Πρέπει να δεχτούμε ένας από τον άλλο, να είμαστε γενναιόδοροι και αν υπάρχει αίσθηση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ε, μία βάση στη συνθήκη, νομίζω μπορούμε να απευθυνθούμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Οπότε εξακολουθούν να ισχύουν κάποιε από τι αρχικές μου σκέψεις. Ε, βεβαίω ο χάρτης είναι χρήσιμος. Βεβαίω η νομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου έχει λάβει υπόψη το χάρτη. Και ο χάρτης βεβαίω είναι 50 ε, χρόνια μετά την ΕΣΔΑ, οπότε είναι πολύ πιο επίκαιρος ε, και βεβαίως αποφελείται και το δικαστήριο του Στρασβούργου από αυτό. Τώρα, ο δικό μου ρόλο θα έλεγα είναι έτσι να είμαι ο επιφυλακτικό, Αντιλαμβάνομαι πω ε, έχει υπάρξει τεράστια πρόοδο στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εθνική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε συνηγόρου του πολίτη, φορεί ίσων δικαιωμάτων, ίσων ευκαιριών και κάνουν ε, βεβαίω θετική δουλειά. Το Equinet, παραδείγματο χάρη, ε, το δίκτυο αυτό των φορέων ισότητας είναι πολύ πολύτιμο μέσο. Έχουμε επίσης αναπτύξει στις χώρες Ένωσης έναν δομημένο διάλογο μεταξύ κρατικών αρχών ακόμα και στο τοπικό επίπεδο και της κοινωνίας των πολιτών και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε λοιπόν τώρα για το τι δεν έχει γίνει ακόμα το μισοάδιο μέρος του ποτηριού ε, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, θεωρώ. Η αντιμετώπιση των Ρωμά, π.χ. στην Ευρώπη, είναι σκανδαλώδης. Έχω ταξιδέψει σε όλες αυτές τις χώρες, μιλάω εκεί πέρα με τους ανθρώπους αυτούς για να καταλάβω πώς βλέπουν αυτή την κατάσταση. Και υπάρχει διάκριση σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. ζουν λιγότερο, γύρω στα 10 χρόνια κατά μέσο όρο, από την πλειοψηφία του πληθυσμού. Τα περισσότερα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο. Σε κάποιες χώρες μόνο τα μισά παιδιά των Ρώμα πηγαίνουν στο σχολείο. Έχουμε επίσης προβλήματα με την απασχόληση, διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σχεδόν κανένας Ρώμα δεν εργάζεται και αυτό είναι πρόβλημα. Κατάσταση της στέγασης, πάρα πολύ άσχημη. Κάποιε από τι κοινότητε αυτές ζουν σε παραγκουπόλεις κατά το οποίο συγκρίνεται με τις φτωχότερε χώρες του κόσμου και, τα, και η πολιτική συμμετοχή τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη στι περισσότερε χώρες. Οπότε υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι. Γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν είχαμε αποτελέσματα. Έχουμε κάνει τόσα συνέδρια, συζητήσεις για την κατάσταση στο όνομά. Είναι λίγες οι αλλαγές επί τόπου. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Δεύτερον, νομίζω πως έχουμε αποτύχει όσον αφορά μια διαδικασία ασύλου και μετανάστευσης που θα πλήρει ορισμένες προδιαγραφές και η συζήτηση αυτή συνεχίζεται. Είναι λυπηρό το ότι η διαδικασία προς μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου απαιτεί τόσο πολύ καιρό. Ελπίζω τώρα να μπορέσουμε να υιοθετηθεί μια τέτοια πολιτική μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Αλλά δεν, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο όταν ακούω τις διάφορες κυβερνήσεις. Το οποίο σημαίνει μεταξύ άλλων πως πολλοί άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και έχουν σοβαρά αιτήματα ασύλου δεν έχουν την ευκαιρία να τα αναπτύξουν. Δεν καταφέρνουν να φτάσουν. Έχουμε μια κατάσταση όπου 2.000 πρόσφυγες ή μετανάστες από την Αφρική πνίγηκαν στη Μεσόγειο φέτος τους τελευταίους 12 μήνες. 2.000 άνθρωποι πνίγηκαν. Πού είναι η αγανάκτηση. μεσογειο φετος τελευταιους 12 μηνες είναι η αλληλεγγύη με αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Που σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν καν το τι συνέβη στους δικούς τους που ήρθαν στην Ευρώπη, πήγαιναν στην Ευρώπη να βγάλουν λεφτά και να βοηθήσουν την οικογένειά τους. Οπότε η Επίτροπο ε, κυρία Μάνεμστρομ εδώ πέρα προσπαθεί να αλλάξει λίγο την ατμόσφαιρα και στις βόρειες χώρες της Ευρώπης και να προσπαθήσει να ζητήσει μια πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών. Και εδώ πέρα φτάνουμε στο τρίτο ζήτημα, ε, την αύξηση της ξενοφοβίας, ε, του ρατσισμού, της λαβοφοβίας και του αντισημιτισμού ακόμα στην Ευρώπη με ακραίες ομάδες που είναι πάρα πολύ δραστήριες ε, όσον αφορά τη δημιουργία ατμόσφαιρας μη ανεκτικότητας και μίσους ακόμα ε, δυστυχώς ε, βλέπετε πράγματα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Ε, έχω απογοητευτεί και σε σχέση με κάποια μίμιε όσον αφορά τις προκαταλήψεις έναντι ευπαθών ομάδων. <coughs> Κατόπιν θεωρώ πως δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τα του οίκου μας όσον αφορά το τι έγινε μετά τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001, η ευρωπαϊκή συμμετοχή στο λεγόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, Καταφέραμε τώρα να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με τον Πολωνό εισαγγελέα που εξετάζει τις κατηγορίες αυτές για τις μυστικές τοποθεσίες στην Πολωνία που βασανίζονταν ύποπτοι. Δεν έχουμε ακόμα τέτοιο διάλογο με τις αρχές της Ρουμανίας αλλά έχουμε στοιχεία για να αποδείξουμε πως και εκεί πέρα είχαμε μια κατάσταση μιας μυστικής τοποθεσίας κράτησης που χρησιμοποιήθηκε για παρόμοιου σκοπούς. Υπήρχαν και άλλες τέτοιες ε, εκδόσεις ε, θα τις λέγαμε. Η δε χώρα μου η Σουηδία δεν έχει ερευνήσει την περίπτωση ε, δύο Αιγυπτίων που παραδόθηκαν στη CIA και μετά πήγαν στο Κάιρο όπου τους βασάνισαν. Εκεί πέρα πρέπει να ξεχαρίσουμε το τι έγινε, Έτοιμα το οποίο έχει έλθει και από δύο φορείς του ΟΗΕ. Οπότε μπορούμε να ασκήσουμε αυτοκριτική, δεν νομίζω πως μπορούμε να είμαστε χαλαροί εδώ πέρα. Βλέπω επίση στον τίτλο του πάνελ αυτού πώς μπορούμε να μιλήσουμε και για το Συμβούλιο της Ευρώπης, άρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ τώρα ως Επίτροπος με απορώ με την καθυστέρηση στη μετάβαση από τον κομμουνισμό σε ένα πιο ελεύθερο σύστημα όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι σε κακή κατάσταση σε πολλές χώρες στην Ευρώπη υπάρχει διαφθορά, πολιτική παρέμβαση και πολλή ανικανότητα. Και αυτό επηρεάζει την ατμόσφαιρα ολόκληρη της χώρας αυτές όσον αφορά την αίσθηση που υπάρχει ε, για τη δικαιοσύνη στις χώρες, κάτι το οποίο μετά έχει και άλλα αποτελέσματα. Οπότε το μήνυμά μου είναι πως το έργο μας δεν έχει τελειώσει παρά την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και τη Συνθήκη της Λισαβόνας και το χάρτη Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα και ανησυχώ να σας πω την αλήθεια για αυτό το οποίο εγώ βλέπω ως μια κρίση αξιών. Όταν μιλάμε για την έλλειψη ανεκτικότητας ε, στις ευπαθείς ομάδες, στους διαφορετικούς και στους όσους έρχονται απ' έξω. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη και φοβούμε πως κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι αξιωματούχοι δεν υψώνουν ε, το ανάστημά τους για να αντιταχθούν σε αυτές τις τάσεις και άρα ε, χωρίς, ε, χωρίς να το θέλουν, χωρίς να είναι σκεμμένο, ε, νομοποιούν την προπαγάνδα, την ακραία στην Ευρώπη και αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Σέζαρ Χέρμα που αντιπροσωπεύει την Πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διευθυντή τη Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Δικαίου του Υπουργείου Εξωτερικών. Κύριε Χέρμα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, που με καλέσατε ως εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου να συμμετέχω μαζί με διακεκριμένους ομιλητές στη σημερινή ακρόαση. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, μετά από την εισήγηση του Επιτρόπου εγώ θα εστιάσω την προσοχή σε θέματα που είναι πιο σημαντικά για τα θεμελιώδη δικαιώματα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έναρξη σε ισχύω του χάρτη μαζί με τη συνθήκη του Λισαβόνας δεν προκάλεσε επανάσταση στα κράτη-μέλη. Όπως γνωρίζουμε, ο χάρτης ισχύει κυρίως ε, στα θεσμικά όργανα και στα σώματα της Ένωσης. Στα κράτη-μέλη ο ρόλος του είναι περιορισμένος για την επιβεβαίωση των δικαιωμάτων αρχών και ελευθεριών που ήδη υπάρχουν στα συντάγματα, γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικέ διεθνεί συμφωνίες. Αυτός είναι ένας από τους λόγους γιατί ο χάρτη ίσως να μην συζητάται τόσο πολύ σε εθνικό επίπεδο όσο στην ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι νομοθεσίε τη Ένωση γενικά είναι εν γέννη σύμμορφε με τον χάρτη. Και αυτό στον ίδιο βαθμό που είναι σύμφωνα, σύμμορφα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλε θεμελιώδει πράξει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγμα που δεν συμβαίνει πάντοτε. Η μη συμμόρφωση, ωστόσο, ακόμα και αν προσδίδει, μάλλον αν προσελκύει μεγάλη προσοχή και ακόμα και είναι σκανδαλώδη, ε, όπω είπε ο Επίτροπο Χάμαρμπεργκ μόλι, είναι εξαίρεση πάντως όσον αφορά τις εθνικές νομοθεσίες και γενικότερα πράξεις εφαρμοστικές. Ωστόσο συμβαίνει και θα πρέπει να τονίσουμε πως τα στεγματικά δικαστήρια των 100 μελών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα έχουν τα κατάλληλα νομικά δεσμευτικά μέσα και μπορούν να βοηθήσουν στην νομιμότητα των, της εθνικής νομοθεσίας και της εφαρμογής της, ώστε αυτή να εμπίπτει στο πεδίο της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό που καθιστά πιο αναγνωρίσιμο το χάρτη είναι μεμονωμένες περιπτώσεις που έρχονται στα ανώτατα εθνικά δικαστήρια ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και οι <clears throat> επακόλουθες αποφάσεις που δηλώνουν ότι μεμονωμένε αποφάσει οι πρακτικέ των εθνικών ε, διοικητικών μηχανισμών παραβιάζουν τι αρχέ του χάρτη. Μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είχε ακόμα αρκετέ ευκαιρίε ώστε να απαντήσει σε γενικές, σημαντικές γενικές ερωτήσεις που προκύπτουν από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του χάρτη. Τα εθνικά δικαστήρια παίζουν πρωτογενή ρόλο στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης και της επιβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν είναι ακόμα αρκετά σίγουρα για το πώς θα πρέπει να εφαρμόσουν το χάρτη, ακόμα και αν ήδη έχουν λάβει καταγγελίες για παραβιάσεις. Η αβεβαιότητα πολλές φορές καταλήγει στην αποτυχία για εφαρμογή των διατάξεων του χάρτη που έχει άμεση ε, ισχύ και επικρατεί της εθνικής νομοθεσίας και επί της δευτερεύουσας νομοθεσίας, δευτερογενούς μάλλον νομοθεσίας της Ένωσης. Επίσης, <clears throat> ισχύει ε, ισχύουν οι γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που όπως αυτές θεσπίζονται από την νομολογία του, δικαστήριου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όπως ο Διευθυντής Πολ Νέμιτς ήδη είπε, οι κατευθυντήριε γραμμέ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με βάση και παραπομπή τη αρχέ αυτέ έχει αυξηθεί και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερε λεπτομέρειε όσον αφορά το νομικό νόημα της νομοθεσίας αυτής, ε, ιδιαίτερα από το δικαστήριο. <coughs> θα πρέπει να αναλύσουμε Κανονικά όλες τις αποφάσεις που περιέχουν οποιαδήποτε παραπομπή στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχει επίσης αβεβαιότητα μεταξύ των ανθρώπων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή του χάρτη. Εδώ συμφωνώ με την παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε στην πρώτη έκθεση για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη το Μάρτιο. Τα περισσότερα ερωτήματα και παράπονα σε σχέση με τη συμμόρφωση προς το χάρτη που παίρνουμε εμεί στο Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν σχετίζονται με τα θέματα εφαρμογής ε, της ε, με τους τομείς μάλλον εφαρμογής της ε, κοινωτικής νομοθεσίας. Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει στα άλλα αλλά σίγουρα επικρατεί μεγάλη σύγχυση για αυτό το θέμα σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη να επικοινωνήσουμε σαφέστερα ώστε να περιορίσουμε το πεδίο των αμφιβολιών. Μια άλλη παρατήρηση της έκθεσης της Κομισιόν που θα ήθελα να αναφέρω είναι ο κατάλογος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αποκαλείται, που θα πρέπει να συνοδεύει κάθε πρόταση της Κομισιόν από την έναρξή της. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γρήγορα αποφάσισαν να μην μείνουν πίσω. Το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του 2010, Δεκεμβρίου 2010 και το Συμβούλιο στα συμπεράσματα του Ιανουαρίου φέτος αναγνωρίζουν ότι τον βασικό τους ρόλο συνομοθέτες για την εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωτών, θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την νομοθετική διαδικασία, καθώς και στις εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το Συμβούλιο τόνισε πως το πλαίσιο αυτό ότι στο πλαίσιο αυτό ακόμα και οι πρωτοβουλίε των κρατών μελών θα πρέπει να σέβονται τον χάρτη. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, όλα τα προπαρασκευαστικά σώματα ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με το Ενωμάδα Εργασίας ΦΡΕΜΠ σε αναπερίπτωση όταν δηλαδή προκύπτουν θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε σχέση με άλλα θέματα που τονίζονται στην έκθεση της Κομισιόν, η Πολωνία εκτίμησε ιδιαίτερα τις ανακοινώσεις της Κομισιόν για νέες προτάσεις όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη που <clears throat> το εγγυάται το άρθρο 47 του χάρτη. Θα ήθελα να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Πολωνική Προεδρία στην νομοθετικά ε, στην νομοθετική εργασία όσον αφορά την πρόταση για οδηγία για τα δικαιώματα στήριξη και προστασία των θυμάτων εγκλημάτων που υποβλήθηκε τον Μάιο. Ένας άλλος τομέας που δεν έχει ακόμα συζητηθεί ούτε έχει εξεταστεί εις βάθος, είναι η εφαρμογή του χάρτη στις εξωτερικές σχέσεις ένωσης. Αναμφίβολα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται από το χάρτη και ως προς αυτή την πτυχή και προκύπτει το ερώτημα του κατά πόσο ο χάρτης ενισχύει τον ηγετικό ρόλο που παίζουν τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω. Και με αυτή τη σύντομη παρατήρηση θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου και σας ευχαριστώ κυρίε και κύριοι για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Χέρμα. Μας παρουσιάσετε τη θέση της Πολωνικής Προεδρίας ότι αφορά την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο ε, εξέφρασε την προθυμία του να αναμίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε στενό διάλογο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και εγώ ως πρόεδρος της δημόσιας αυτής ακρόασης σας εθαρρύνω να διαβιβάσετε στο Συμβούλιο την ανάγκη εφαρμογής και εμπράκτος αυτής της δέσμευσης που έλαβε για στενότερο διάλογο και συνεργασία με το Συμβούλιο. Τώρα θα καλωσορίσω ένα μέλο όχι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, την κυρία Κέρστιν Λάντγκριν, που είναι η για την έκθεση που αφορά τον αντίκτυπο τη συνθήκη Λισαβόνα στα θεμελιώδη δικαιώματα. Εκπροσωπεί το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Καλωσορίστε, κυρία Λάντγκριν, και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Thank you for having this uh, seminar ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στο σεμινάριό σας. Όπως είπατε, είμαι η συγγήτρια της αντίστοιχης έκθεσης για τη συνθήκη της Λισαβόνας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις αξίες. Παρόλο που υπάρχει κρίση αξιών αυτή τη στιγμή, διαπιστώνουμε ότι η Σύνθηκη της Λισαβόνας και το Συμβούλιο της Ευρώπης εδράζονται στις ίδιες αξίες, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο αυξανόμενος ρόλος, ενισχυμένος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παραδοσιακούς τομείς δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως είναι ε, ο τίτλος Επιτροπής σας, πολιτικές ελευθερίες, ελευθερία, ασφάλεια, ε, πειράζει τα κράτη-μέλη στις διαπραγματεύσεις της νέας σύμβασης, της νέας συνθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στους τομείς αυτούς. Όπως είπα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, το λέω και στην έκθεσή μου, αποτελεί το γνώμονα, το συγκριτικό κανόνα για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη. Και θέλουμε να εφαρμόσουμε πλήρως αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται και από την Επιτροπή σα και από όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Ω Κοινοβουλευτική Συνέλευση ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης καλωσορίζουμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου του 2010. Εκεί ταχθήκατε υπέρ της ε, προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το χαρακτηρίσατε ως ε, θεμελιώδες ε, πρώτο βήμα που θα συμπληρωθεί με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες ε, συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επικροτούμε και το επικοδομητικό πνεύμα με το οποίο οι εκπρόσωποι των θεσμικών μας οργάνων κατέληξαν σε συμφωνίες για πολλά θέματα όπως η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σώματα που ε, εκλέγουν τους δικαστές ε, στο, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έγιναν διαβουλεύσεις και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ευελπιστούμε ότι, και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε μάλλον ότι τέτοιες ε, διαβουλεύσεις θα γίνουν και στις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις για διάφορες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε συνεργασία μαζί σας για να αφυπνίσουμε καλύτερα το κοινό και να προωθήσουμε την προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ Συμβουλίου της Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη θέση τη της Συνθήκης Λισαβόνας θα εξασφαλίσει ε, συνοχή μεταξύ του πανευρωπαϊκού σχεδίου που προωθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης και της διαδικασίας ολοκλήρωσης που εγγενίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα καταλήξουμε τελικά σε ένα κοινό χώρο για προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, κάτι που εξυπηρετεί όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προσχώρηση στην ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και σε άλλες ε, συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης και τους αντίστοιχους ε, μηχανισμούς παρακολούθησης. Έχω ένα όνειρο Το όνειρό μου είναι να συμφωνήσει και η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ώστε να διαμορφώσουμε ένα πανευρωπαϊκό χώρο ελαχίστων προδιαγραφών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δύο είναι οι δρόμοι που μπορεί να μας οδηγήσουν στην υλοποίηση αυτού του ονείρου. Καταρχήν η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεύτερον μια συνολική εναρμόνιση των κανόνων και των προδιαγραφών και της αξιολόγησης των προδιαγραφών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά είναι το κλειδί. 47 κυβερνήσεις και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα ε, 27 κυβερνήσει και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα θα υπακούν στους ίδιους κανόνες και προδιαγραφές και θα ελέγχονται από το ίδιο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έτσι, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χαίρουν αντίστοιχες προστασίες ε, και δικαιωμάτων κατά των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που ήδη ισχύει στα μέλη που έχουν προσχωρήσει στο Συμβούλιο της, ε, στη Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης ε, θα υπάρξει ένα εξωτερικό έλεγχο ε, στο νομικό σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. θα βελτιωθεί η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δέσμευσή της εντό και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προ την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Βέβαια υπάρχει και η αδύρυτη ανάγκη ανανεωμένης πολιτικής δέσμευσης ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, γι' αυτό και θα πρέπει να αναλυθεί νέα δέσμευση από τα διάφορα πολιτικά όργανα, προκειμένου να υποστηριχθεί και να υλοποιηθεί αυτή η προσχώρηση, η ένταξη. Και αυτή είναι πραγματικά μια κρίσιμη στιγμή, στιγμή που διανύουμε. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, ο καθένας στο επίπεδό του για να πραγματοποιηθεί αυτή η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα, συνοχή των διαφόρων προδιαγραφών και εφαρμογή και αξιολόγηση των προδιαγραφών. Χάρη στην προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάφορες συμβάσεις και συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουμε όμως και άλλες προκλήσεις σήμερα. Και υπάρχει δυνατότητα θέσπιση και νέων συμβάσεων για παράδειγμα, σύμβαση, συνθήκε για την προστασία του το εγκλήματο στον κυβερνοχώρο, προστασία δεδομένων, σωματεμπορία, πρόληψη, προστασία από τρομοκρατικέ ενέργειε, αλλά και προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε μηχανισμό παρακολούθηση. Και θα πρέπει να αποφύγουμε και επικαλύψεις και κακή χρήση των κονδυλίων, των, των χρημάτων των φορολογουμένων. Και επίσης αποφύγουμε την κόποση από υπερβολική παρακολούθηση αυτής της εφαρμογής. Ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να έχουμε συστηματικές και ανοιχτές διαβουλεύσεις μεταξύ των ε, οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης και των κοινοτικών οργάνων καθ' όλη τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και ιδιαίτερα στα πλαίσια των νέων νομοθετικών πρωτοβουλειών. Έτσι θα αποφύγουμε τις επικαλύψεις και θα αποφύγουμε και την ε, ε, υποβάθμιση των προδιαγραφών. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε και να ενισχύσουμε την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σε καμία περίπτωση να μην ε, αποδυναμώσουμε τις προδιαγραφές. Όπως είπε πριν από λίγο και ο Επίτροπος Χάμαρμπερκ, Ελπίζω να μην έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ μας. Να μην κάνουμε ε, αγώνα ποιος θα έχει το περισσότερο κύρος και την περισσότερη έγλη. Με κοινές προσπάθειες θα διαμορφώσουμε ένα πανευρωπαϊκό χώρο για, τις βασικές, για τη βασική προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων προς όφελος των πολιτών μας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια δεν θα δημιουργήσουμε νέε τάξεις, ε, νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σε μία περίοδο οικονομικής και πολιτικής κρίσης θα παρουσιάσουμε ένα κοινό πανευρωπαϊκό σχέδιο που θα σέβεται, προωθεί και θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό θα το κάνουν όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και της Ευρώπης από, από όπου και όπου εκπορεύονται. Σας ευχαριστούμε κυρία Λάνγκριν, σας ευχαριστούμε που ήρθατε στη δημόσια ακρόαση. Όπως είπε η συγκεκριά μας στην αρχή της ακρόασης, χαιρόμαστε γιατί ε, συμμετέχουν στην ακρόασή μας και πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και έτσι θα μας πούν από πρώτο χέρι τις εμπειρίες τους από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τελευταίος ομιλητής του πρώτου μέρους της δημόσιας ακρόασης είναι ο κύριος Νίκολας Μπέγκερ, στον οποίο θα δώσω και το λόγο. Είναι διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκών ε, Θεσμικών Οργάνων της Διεθνούς Αμνηστίας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές. Ονομάζομαι Νίκολα Μπίκερ και είμαι διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας της Βρυξέλλας, αλλά επίσης μιλώ εξ ονόματος ε, της ανησυχίας περίπου 100 ε, ΜΚΟ που είναι μέλη του δικτύου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της κοινωνικής πλατφόρμας και ανησυχούν όσον αφορά τη δράση της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της Ένωσης ε, είμαι ευτυχής που γίνεται αυτή η ακρόαση και που βρίσκομαι δίπλα σε τόσο διακεκριμένους ε, εκπροσώπους και φορείς. Πριν δύο χρόνια μέσα σε μεγάλους πανηγυρισμούς παρουσιάστηκε ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η έναρξη μιας εποχής, ε, μιας νέας εποχής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν από ένα μήνα μόλις όμως αυτό το κοινοβούλιο μαζί με την Επιτροπή και την Επιτροπή Αναφορών του ίδιου του Κοινοβουλίου κάναμε ένα σεμινάριο όσον αφορά την αναδίπλωση Μάλλον, ε, σχετικά μάλλον με τη χρήση του χάρτη για την αντιμετώπιση των παραπώνων των πολιτών. Οι φιλοδοξίε της Ένωσης φαίνεται κάπου να λοξοδρόμησαν στα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό που θέλει τώρα η Ένωση είναι μια επιθυμία να διαλύσει τις ε, παρεξηγήσεις για το πού και πότε ισχύει ε, αυτός ο χάρτης, να αποφύγει το να απογοητευτούν οι υπόλοιποι πολίτες. Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι αυτό είναι κάπως, ε, μας θυμίζει κάπως καταστάσεις Κάφκα. τα ανθρώπινα δικαιώματα περνούν κρίση στην Ευρώπη και δεν είναι κάτι το καινούριο. Ήδη έχει χτυπήσει και ο Τόμας ε, μας περιέγραψε πολύ ωραία το τι συμβαίνει και ο κόσμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρεξήγησε τον χάρτη, πολύ καλά τον κατάλαβε μάλιστα. Σας διαβεβαιώ λοιπόν πως τα ανθρωπίνα δικαιώματα θα συνεχίσουν να χτυπούν στην πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τελευταία χρόνια το μέλη του Ευρωκοινοβουλίου έχουν δώσει σαφές μήνυμα. 60% των περιφερειών τους σας θέλουν να εστιάσετε στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διπλάσιο ποσοστό από ό,τι για τα υπόλοιπα θέματα. Εσεί οι Ευρωβουλευτέ είστε έτοιμοι να αναλάβετε αυτή την πρόσκληση. Και ποια είναι η απογοήτευση που φοβάται η Κομισιόν. Πολλά υπόθηκαν πρόσφατα για το αντίφαση ανάμεσα στη δημοσιότητα που δόθηκε για το ξεκίνημα του, ανθρωπίνου, του χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ε, αποκλιμάκωσης. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όταν εμείς ε, θίγουμε ε, υποθέσεις όπως ας πούμε η Ρωμά που δέχονται επιθέσεις στην Ουγγαρία και την Βουλγαρία, ξεχως, ε, ξενοφοβία, κρυφ, ε, συγκαλυμμένες φυλακές τη CIA κτλ. Η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Πολύ άσχημο αυτό, πραγματικά λυπούμεθα που το ακούμε, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Ένωση. Βασικά μας λένε δηλαδή ότι ο χάρτης, αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικός, στην πραγματικότητα είναι ε, άχρηστος, γιατί δεν φέρει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Ποια είναι η παρεξήγηση λοιπόν αυτή και πώς συνέβη. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο λυπηρό. Το άρθρο 51 του χάρτη είναι αυτό που παρατίθεται πιο συχνά, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύουν κανέναν. Είναι αυτό που περιορίζει τα δικαιώματά μας. Το άρθρο 51 λέει πως ο χάρτης ισχύει μόνο εντός ε, της εντολής της Ευρωπαϊκής ε, Κοινότητας και στα κράτη-μέλη μόνο στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν επιφέρει καμία νέα εξουσία ή αρμοδιότητα στην Ένωση. Τα δεχόμαστε όλα αυτά, ναι, μεν, και μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεμένα τα χέρια της και ότι διστάζουν τα κράτη-μέλη να δουν και το δικό τους, ε, το το πώς τα καταφέρουν και δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό ούτε για τώρα, ούτε για το μέλλον, δυστυχώς. Κατά κάποιο τρόπο ο χάρτης αυτός έχει περιορίσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, για τις καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς ε, αυτή είναι η παρεξήγηση, πρέπει να πούμε στις Επιτρόπους Μάλστρομ. <coughs> Ακόμα και αυτοί που το χρησιμοποιούν ε, μάλλον σε διαρκώς ακούμε αυτή τη δικαιολογία ότι όπου το παρεξηγήσατε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χάρτη. Οι περισσότερες ΜΚΟ πιστεύουν πως χρησιμοποιείται ο χάρτης ωστόσο για ακριβώς να επιτίθεται ενάντια των ε, αξιών που υποτίθεται πρέπει να προωθεί. Ο χάρτης ε, συντάχθηκε όχι μόνο πριν από δύο χρόνια, πριν από 12 χρόνια και όπως ακούσαμε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στα εθνικά ε, δικαστήρια και στα, και στα κοινοτικά την τελευταία δεκαετία. Η φύση όμως των δικαιωμάτων αποτελεί μια οντότητα και θα πρέπει να αποκτήσει σάρκα και οστά καθώς προχωράμε. Εστιάζοντας λοιπόν στο άρθρο 51, καταστρέφουμε αυτό το ζωντανό σώμα, αυτή την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Και αυτό που είναι περίεργο είναι ότι αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει τις αρμοδιότητες που χρειάζεται για να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το έχει αυτό σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Ούτε ο χάρτης ούτε οι συνθήκες λείπουν. Χτυπάμε λοιπόν στη σωστή, στην κατάλληλη πόρτα. Το μήνυμα μας στην Ένωση είναι σαφές. Μην περιορίζετε τις αρμοδιότητες που ήδη έχετε. Να σας δώσω τρία παραδείγματα όπου κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβαίνει για τις διακρίσεις. Αυτή η αρχή περιλαμβάνεται στο χάρτη και στις ε, συνθήκες της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οθετήσει δεσμευτικά όργανα εδώ, όπως για παράδειγμα την ε, οδηγία περιφυλής που απαγορεύει τις διακρίσεις που βασίζονται στην θεωτική προέλευση. Γιατί λοιπόν δεν ενεργεί όταν ας πούμε παράνομα αναφέρονται οι Ρωμά. Πρέπει να επεκταθεί ώστε να ε, καλύπτει τις περιοχές που καλύπτουν οι συνθήκες Δείτε τις περιπτώσεις του ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις αρμοδιότητες που χρειάζεται. Νέες νομοθεσίες και οι κρατικέ επίσης νομοθεσίες ισχύουν. Ισχύει ο χάρτης σε όλα αυτά. Γιορτάστηκε το γεγονός ότι περιλαμβανόταν το άσυλο σε αυτό το χάρτη. Τι εμποδίζει λοιπόν την Ένωση από το να το εφαρμόσει. Έλλειψη ελέγχου και λογοδοσίες και συνενοχή στις, στις ε, φυλακές της CIA, τις μυστικές φυλακές της CIA. Και εδώ τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να ερευνήσουν την κατάσταση. Τίποτα ωστόσο δεν αναφέρεται για το τμήμα του χάρτη, ότι απαγορεύονται δηλαδή τα βασανιστήρια. Δεν είναι πια αυτό δηλαδή τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απαγόρευση των ε, ε, βασανιστήριων. Πιστεύουμε πως ε, έχει δημιουργηθεί μια σαλμένη αντίληψη. δεν είναι το πρόβλημα το 51 το πρόβλημα. Είναι το ότι δεν χρησιμοποιούμε το άρθρο 7 τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει πολιτικό μηχανισμό ώστε να προλάβει σοβαλέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό μόνο θεωρείται επιλογή. Αυτό οδηγεί στο άρθρο 2 που αναφέρει όλες τις αξίες και τα δικαιώματα από τα οποία αναφέρονται εδώ, κάτι τα οποία δεν είναι εφαρμόσιμο. Εμείς πιστεύουμε πως το άρθρο 2 και το 7 χορηγούν στα θεσμικά όργανα την ε, αρμοδιότητα να αξιολογήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Και το άρθρο 7 δεν αφορά την ταπείνωση των κρατών μελών. Δεν θέλει να κάνει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση χωροφύλακα, αλλά βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξει κατά πόσο τα κράτη-μέλη σέβονται αυτά που έχουν αναλάβει να κάνουν μέσω όλων των συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν συνυπογράψει. Και εσείς που έχετε το δικαίωμα πρωτοβουλίας χρησιμοποιήστε το να σταματήσετε πια να αγνοείτε αυτή την κατάσταση. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν χρειάζεται να επανεφεύρουν τον τροχό ή να αποκτήσουν ε, εξαιρετικές νέες αρμοδιότητες. Ε, έχετε αρμοδιότητες και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε και τις ε, αρμοδιότητες που έχουμε δώσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στους μηχανισμούς εποπτείας του να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά τον Ρώμα τώρα. Μπορείτε να σταματήσετε την κατάσταση των τον άσυλο να πάψουν να ζουν σαν να είναι υπάνθρωποι. Να μην χρησιμοποιούμε δικαιολογίε πλέον. Είναι πλέον καιρός να είμαστε έντιμοι με του εαυτούς μας για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ο καιρό των ε, προσχημάτων και των δικαιολογιών έχει περάσει προπολού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τις νομικές του εξουσίε, αρμοδιότητες και όχι πια μόνο λόγια. Μπορούμε να βασιστούμε σε εσά. Ελπίζω πως ναι. Ε, Ευχαριστώ. Τώρα ξεκινήσει η συζήτηση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως για να μπορέσουμε να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις θα περιοριστεί ε, ο χρόνος ομιλίας σε δύο λεπτά αναπαρέμβαση. Οπότε, όσοι θέλουν τώρα να παρέμβουν, όπως ανέφερα στην αρχή, δεν θέλουμε να ακούσουμε ευρωβουλευτές μόνο. Οπότε μπορείτε να μας δώσετε τα ονόματα σε ένα χαρτί, θα το μαζέψει η γραμματεία. Ή όταν σηκώνετε το χέρι σας ε, να συστήνεστε. Gomez. Κυρία Γκόμες, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μα δεν είναι ηρωνικό ότι τη στιγμή κατά την οποία οι πολίτες μας θεωρούν πως όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και η δημοκρατία παραβιάζεται από αυτούς που υποτίθεται πως ε, την ε, ε, διαφυλάττουν εντός ενός και μιλάω εδώ πέρα για το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω πως το πρόβλημα είναι και εντός ε, του Κοινοβουλίου και χαίρομαι για το ότι πράγματι απευθυνθήκατε στο Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσετε τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, αλλά στο Κοινοβούλιο βλέπουμε κάτι το ενδιαφέρον. Έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα στο εξωτερικό και θεμελιώδη δικαιώματα στο εσωτερικό. Είναι αρνητικό Δηλαδή σαν να μην ισχύουν τα ίδια πράγματα. Και θα ήθελα να πω πως να ζητήσω τον κύριο Μπέγκε αν μπορεί να μας πει τι άποψη έχει για την έλλειψη λογοδοσίας για τη CIA και τις παραδόσεις εκείνες. Γιατί επειδή οι κυβερνήσεις όλων των πολιτικών αποχρώσεων και της δικής μου οικογένεια είναι συνένοχες και δεν θέλουν να δώσουν λόγο. Και αυτό φαίνεται και στην αδράνεια του Κοινοβουλίου. E αυτό έχει συνέπειες για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρείται αξιόπιστη. Και όταν έρχεται σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη εγγύηση εξωτερικού αν θέλετε οπότε ήθελα να σε ρωτήσω πώς το βλέπετε εσείς αυτό ευχαριστώ κύριε Σκολιά ευχαριστώ πιστεύω ότι όπως είπαν και πολλοί προλαλήσαντες, mm -hmm. πολλοί προσκεκλημένοι, ε, ο χάρτης είναι ένα βήμα πρόοδο αλλά δεν αρκεί αυτό. Συμφωνώ. Και μου άρεσε και η ομολογία του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είπε ότι ήταν αρχικά επιφυλακτικό, σκεπτικιστής απέναντι στο χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων, αλλά τελικά μεταπίστηκε. Και υπάρχει όντως μια διαφορά μεταξύ του γράμματος του νόμου και της εφαρμογής αυτού του γράμματος. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς αυτή τη διαφορά. Ακούσαμε τι είπε η κυρία Γκόμες, ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί περίτρινη απόδειξη αυτής της διαφοράς. Μερικοί αναφέρθηκαν στην, στις παράνομες δραστηριότητες CIA στην Ευρώπη. Ο κύριος Σάμερμπερκ μίλησε εκτενώς γι' αυτό και, συγγνώμη, και πέρασε ένας χρόνος μέχρι να αναλυθεί η πρωτοβουλία ε, να γίνει στην Επιτροπή ΛΙΜΠΕ μία αξιολόγηση των, της αποτελεσματικότητας των συστάσεων και των ψηφισμάτων που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό, Κοινοβουλίο, ε, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Οπότε δεν ήταν αρκετά γρήγορο, ούτε αρκετά επιμελές ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρακολουθήσει την ε, έμπρακτη εφαρμογή των προτάσεων που είχε κάνει με δική του πρωτοβουλία, ώστε να στιγματιστούν αυτές οι παράνομες δραστηριότητες της CIA στην Ευρώπη. Το πιο σημαντικό όμως ε, είναι να ε, ατενίζουμε το μέλλον και να μην ασχολούμαστε μόνο με επικριτική αξιολόγηση του παρελθόντος. Πολλά έχουν γίνει στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα θεμελιώδη δικαιώματα ποιες είναι οι συστάσεις των προσκεκλημένων μας προκειμένου ε, να βελτιώσουμε και να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστούμε, Κάρλος. Κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους προσκεκλημένους και ιδιαίτερα τους κυρίους Χάμαμπερκ και Μπέγκερ για την ε, κριτική στάση τους απέναντι στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Και να θέσω και μία ερώτηση στην Πρόεδρο ή στους Συμπρόεδρους. Προσκαλέσαμε τις Επιτρόπους Ρέντινγκ και η Μάλμστρομ. Και δεν ήρθαν ή δεν τις προσκαλέσαμε καν. Καλό θα ήταν να, να το και οι δύο Επίτροποι. Γιατί είναι χρήσιμο το έργο τους και μακάρι να ήταν εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμώ σε καμία περίπτωση ...τη παρουσία και θέση του κυρίου Νέμιτς αλλά νομίζω ότι οι επίτροποι εκπροσωπούν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, την εκπροσωπούν και προς τα έξω. Έχω μία ερώτηση προς τον Επίτροπο Χάμαρμπερκ για τη σχέση της σύμβασης, ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του θεμελιώδη χάρτη, ε, του χάρτη θεμελιώδων δικαιωμάτων. Όπως είπατε, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι πάνω από 50 χρονών θεσπίστηκε αμέσω μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ ο χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων είναι κάτι καινούριο και περιλαμβάνει διατάξει που την εποχή σύνταξη τη Ευρωπαϊκή σύνταξη ήταν αδιανόητε. Για παράδειγμα, η πάταξη διακριτική μεταχείρισης για ε, λόγου γενετήσου προσανατολισμού. Τότε ήταν αδιανόητο να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Σήμερα υπάρχει και σχετική διάταξη για προστασία. Επίση, υπάρχει μερικέ φορέ σύγχυση, το επισημάνετε και εσεί, κυρία Λάντγκριν, μεταξύ των δύο εργαλείων, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μήπως λοιπόν θα μπορούσατε να μας πείτε πώς πιστεύετε ε, πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιο συχνά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Αναφερθήκατε στη νομοθεσία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ουγγαρία. Ε, με δυσαρέστησε αυτή η πληροφορία, γιατί και εμείς αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περίμεναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο κατηγορηματική απέναντι στην Ουγγαρία και πιο αυστηρή ε, για τον νόμο αυτό για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και περιμένουμε στενότερη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συχνή προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα μας εξυπηρετούσε και εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι τέτοιο. Όσο μιλούσατε, ιδιαίτερα όσο μιλούσε ο κ. Μπέγκερ, σκεφτόμουν το εξής. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε ε, να παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίε, την πιέζουμε και θέλουμε και στενή συνεργασία μαζί της. Αλλά τα προβλήματα κυρίω τα αντιμετωπίζουμε στη σχέση με το Συμβούλιο, με τα κράτη-μέλη. Και το ίδιο είχαμε και με, τον νόμο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ουγγαρία και πριν από δύο χρόνια όταν ε, θελήσαμε να καταρτήσουμε το ψήφισμα για τη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, ε, επευκαιρία της Ιταλικής περίπτωσης και τελικά δεν συγκεντρώσαμε την πλειοψηφία που χρειαζόμασταν και δεν πέρασε το ψήφισμα. Είναι δύσκολο μερικές φορές και αυτό. Και κάτι άλλο, μια δήλωση περισσότερο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαρτάται από την κοινωνία των πολιτών και περιμένει όχι μόνο ενημέρωση και πληροφορίε, αλλά και πίεση προ εμά, αλλά και κυρίω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Θέλουμε οι ακτιβιστέ και οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών να διεκδικούν και να απαιτούν την εφαρμογή και την άσκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εμείς θεωρητικά κατοχυρώνουμε. Ευχαριστούμε κυρία Λούνατσεκ. Θα ήθελα να θερμοπαρακαλέσω τους συναδέλφους να μην ξεπέρνουν το δίλεπτο στις ε, παρατηρήσεις του, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις του πάνελ. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το κατά πόσο προσκαλέσαμε και τις Επιτρόπους. Η γραμματεία μου είπε ότι προσκαλέσαμε και τις δύο Επιτρόπους, Ρέντινγκ και Μάλμστρομ. Η κυρία Μάλμστρομ αρνήθηκε την πρόσκληση λέγοντας ότι δεν είναι δική της ευθύνη, είναι ευθύνη της κυρίας Ρέντινγκ και η κυρία Ρέντινγκ είχε ενηλυμένες υποχρεώσεις για σήμερα το απόγευμα. Οπότε, γι' αυτό μας έστειλαν τον Γενικό Διευθυντή τον αρμόδιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Λάτφορτ. Um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτηση που θα έκανα ήδη ακούστηκε από τον κύριο Κοέλιο. Δηλαδή τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης για να συνεργαστούν στο μέλλον. Οπότε θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Νομίζω πως είναι θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, ενταχθεί και εκείνη στην σύμβαση γιατί έτσι θα ολοκληρωθεί, θα κλείσει ένας κύκλος και νομίζω πως έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε την αμηχανία και τη ζήλια αν θέλετε που υπήρχε για να λειτουργήσει το σύστημα. Γιατί είχαμε το παράδοξο πως ο Τόμας Χάμαρμπεργκ, ο οποίος δραστηριοποιείται ε, ενεργά έχει λιγότερη εξουσία, ενώ η δική μας η Επίτροπος έχει περισσότερη, περισσότερες αρμοδιότητες, δηλαδή πιθανές κυρώσεις, αλλά είναι απρόθυμη να τις χρησιμοποιήσει. Εκεί κάπου υπάρχει η δυνατότητα για να κάνουμε μια κυκλωτική κίνηση, αν θέλετε, και να χρησιμοποιήσουμε και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πείσουμε τα πρόθυμα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν. Πρέπει και εμείς βεβαίως να δούμε τι νομικές διεξόδους ε, έχουμε που δεν είναι βεβαίως τόσο εκτεταμένες ε, όσο αυτές της Κομισιόν ή του Συμβουλίου. Θα το δούμε αυτό άλλη φορά. Αλλά το βασικό πρόβλημα νομίζω που ανέφερε και η Ουλρίκα Λούνατσεκ εντό του Κοινοβουλίου είναι αυτή η απροθυμία ότι κάποιοι με βάση εθνικούς λόγους λένε δεν θέμε να μας ελέγχεται. Ως αν είμαστε μια διπλωματική λέσχη. Δεν είμαστε μια διπλωματική λέσχη, είμαστε μια κοινότητα δικαίου. Και έχουμε συμβατικές υποχρεώσεις και ε, υποτίθεται πως αυτό ακριβώς είναι η δύναμή μας, ότι μπορούμε ο ένας να ελέγχουμε τον άλλον, γιατί ειδικά στον τομέα του ποινικού δικαίου, αλλά συνολικά στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασιζόμαστε στην αμοιβαία εφαρμογή και σεβασμό των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει σύμφωνα με την συνθήκη και την ε, σύμβαση. Οπότε όλο αυτό το οικοδόμημα στηρίζεται, σε αυτό το επίπεδο μας στηρίζει το ένα στον άλλον. Οπότε το ότι συμβαίνει σε μια χώρα έχει σημασία σε άλλη. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν τομεί ταμπού. Υπάρχουν προβλήματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση και να ξεπεράσουμε αυτές τις αναστολές. Ευχαριστούμε Σάρα. Τελευταία παρέμβαση. Η κυρία Εξανθιά εκεί στο βάθος, δεν σας ξέρω. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ονομάζομαι Μαριφέ Φιλερινού. Από την ΜΚΟ καταγγελία των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο τα όσα αναφέρθηκαν από τον κύριο Χαμαρμπέργκα νομίζω ότι βασικά οφείλονται στην ακραία φτώχεια. Πώς η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας ως ε, ανθρωπίνου δικαιώματο, θεμελιώδου ανθρωπίνου δικαιώματος μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω πως αυτό θα πρέπει να εντάσσεται απόλυτα το θέμα της ακραίας στόχιας στις προτεραιότητες του Οργανισμού Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε αυτά να μπορούν να αντιμετωπίζονται σε συγκεκριμένου τομεί, στον τομέα τη απασχόληση, του πολιτισμού, της παιδεία, της υγεία, της δικαιοσύνη, τη προστασία τη οικογένεια και του ε, παιδιού. της κατάρτισης και νομίζω πως ε, στο επόμενο πολιετές πρόγραμμα θα πρέπει αυτά τα θέματα να εμφανίζονται ρητά. δεύτερο θέμα αφορά τις διακρίσεις κοινωνικού προέλευσης. Τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας στόχια, υπόκεινται σε διάφορες διακρίσεις κοινωνικής φύσης, όπου είναι στο άρθρο του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά ποτέ δεν αναφέρεται. Πρέπει πλέον αυτές, αυτή η διάκριση κοινωνικής προέλευσης να θεωρηθεί επίσης απαράδεκτη και παράνομη μέσω του οργανισμού αλλά και με άλλα μέσα. Να πω επίσης ότι συμφωνώ με την παρατήρηση του Νικολά Μπέγκερ ότι δεν μπορούμε να απαντούμε στους ανθρώπους που είναι που ζουν στη φτώχεια, ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ένα στόχο κατά πολέμηση τη φτώχεια. Και θα πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτού του στόχου όσον αφορά την πραγματική πρόσβαση στα, ανθρώπινα στα θεμελιώδη δικαιώματα. Και τέλο, η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορούμε να μιλάμε παρά για την υπογραφή του, του, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και για την ε, προσυπογραφή του θεμελιώδους χάρτη. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Νέμιτς, μετά στον κύριο Χάμαρμπεργκ και θα ρωτήσω και τον κύριο Χέρμαν θέλει να παρέμβει, όχι. Έπειτα η κυρία, ο κύριος Μπέργκερ και η κυρία Λούντγκρεν. Ο κύριος Νέμιτς πρώτος. Um, Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει πολύ στα σοβαρά την υποχρέωση της να είναι θεματοφύλακα στις συνθήκες του κοινοτικού δικαίου αλλά και του χάρτη θεμελιώδων δικαιωμάτων και αυτή η ευθύνη προϋποθέτει ότι όταν ασκούμε προσφυγή στο ΔΕΚ να έχουμε μεγάλη βεβαιότητα ότι θα κερδίσουμε γιατί κάθε υπόθεση που χάνουμε στο ΔΕΚ υπονομεύει τη θέση και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μελλοντικές προσφυγές και υποθέσεις πολλά άκουσα σήμερα, αλλά το κράτος δικαίου, πέραν των διαφωνιών, σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί ε, στις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα. Γιατί αν κάποιος θεωρεί ότι έχει νομικές δυνατότητες που δεν έχει, αυτό δεν είναι προς του πολίτη από αυτή την άποψη θα αναλάβει τις ευθύνες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα και πολλές δηλώσεις σήμερα που είναι ακριβείς. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις παράνομες προσαγωγές κρατουμένων. Όλοι οι επίτροποι που ήταν αρμόδιοι σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων έλαβαν δράση και ανέλαβαν δράση και είχαν διάλογο με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και μάλιστα και με επιτυχία. Έχω για παράδειγμα την περίπτωση της Πολωνίας. Εκεί ξεκίνησαν διώξεις το ανέφερε και ο κύριος Χάμαρμπεργκ. Και αυτό έχει σχέση και με την ε, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει, είναι χάρη και στην συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια αυτά δεν προβάλλονται για προφανείς λόγους πάντα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι αυτό το θέμα δεν εμπίπτει αυστηρά στις νομικές μας αρμοδιότητες, αλλά σίγουρα ε, δεν ε, είμαστε αμέτωχοι. Ε, λαμβάνουμε ό,τι πρωτοβουλίες μπορούμε στα πλαίσια και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να πω και δύο λόγια για τα επιμέρους ζητήματα που υπέβαλε ο κύριος Χάμαρμπερκ. Θα μπορούσα και εγώ να ασχοληθώ με τα ίδια θέματα και να υπογραμμίσω τις δράσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους Ρωμά για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε πολύ σοβαρά υπόψη την πιθανότητα άσκησης νομικής προσφυγής και μάλιστα κατέπτυσε και ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει αυτό το στοιχείο της παιδείας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, των κοινωνικών ζητημάτων που επισημάνατε. Έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των δικαιωμάτων, όχι νομικιστική. Και η ανακοίνωση για τους Ρωμά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης μας. Στην τελευταία παρέμβαση για τα κοινωνικά δικαιώματα και το χάρτη, το χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων, ε, θα ήθελα να πω ότι επί της ουσίας συμφωνούμε. Αλλά έχουμε οργανισμό αρμόδιο με συγκεκριμένη εντολή να παρακολουθεί την εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων, ακόμη και την περίπτωση κοινωνικής, κοινωνικών διακρίσεων, πρόσβαση, περιορισμό της πρόσβασης α, ατόμων από φτωχές οικογένειες σε παιδεία, στην παιδεία ή σε άλλες ευκαιρίες που δίνουν οι κοινωνίες και το θέμα των βιωτικών συνθήκων. Θέλουμε απλώς να αποφύγουμε και την επικάλυψη, το ανέφερε και εκπρόσωπο Συμβουλίου της Ευρώπης δεν μας συμφέρουν διπλές εντολές και επικαλύψεις σε οργανισμούς που ούτως ή άλλως είναι εν μέρει ανεξάρτητοι. Και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφεύγει την ε, ανάθεση ε, παρόμοιων εντολών ή εντολών που επικαλύπτονται. Γιατί πραγματικά, αν έχουμε τέτοια επικάλυψη εντολών, πραγματικά θα κατακασπαταλούμε τα κοινοτικά κονδύλια, που ούτως ή άλλως είναι σπάνια. Θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοια διασπάθηση των πόρων. Το θέμα και τη σύμβαση είναι πολύ σημαντικό που γίνεται, και γίνεται και μεταξύ των του Προέδρου του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Προέδρου του ΔΕΚ, αλλά και με Προέδρους των Συνταγματικών Δικαστηρίων των Κρατών Μελών. Και ανακύπτει η πρόταση για μια πολυεπίπεδη συνεργασία. Η συνεργασία αυτή προσπαθεί να καλύψει όλα τα μέτωπα προκειμένου να αποφευθούν και τα κενά αλλά και οι επικαλύψεις με στόχο την πλήρη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Βέβαια αυτό το θέμα είναι πολύ σύνθετο, περίπλοκο και σίγουρα το Ευρωβαρόμετρο δεν θα σας δείξει πλήρη συμφωνία γιατί στην δημοκρατία έχουμε πολλές πτυχές και δεν φαίνονται πάντα κάτι αυτές αλλά θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την πολυμορφία, την περιπλοκότητα, να τη διαχειριστούμε σωστά για να εξυπηρετήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Και θα πρέπει να εμπνευστούμε από αυτό το διάλογο που έχουν οι δικαστικές αρχές και να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο, στο διάλογο των εκτελεστικών εξουσιών, στο διάλογο των διοικήσεων, των διαφόρων σωμάτων, ώστε να έχουμε παρόμοια, παρόμοιο πνεύμα συνεργασίας πολυεπίπεδο να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο δίκτυο ώστε ένας πολίτης που διαμαρτύρεται να καθοδηγείται προς το αρμόδιο όργανο που θα μπορέσει πραγματικά να τον βοηθήσει και να μην τον στέλνουμε από τον Άννα στον Καϊάφα. Πάντως συμφωνώ ότι η πρακτική, η έμπρακτη εφαρμογή του νόμου είναι εξίσου σημαντική με το γράμμα του νόμου. Σημείωσα και τις ε, επικρίσεις και τις κριτικές παρατηρήσεις που διατυπώσατε. Πάντως το σημαντικό για το νόμο και για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι να λαμβάνουμε αυτό το θέμα σοβαρά υπόψη και να το χειριζόμαστε με αξιοπρέπεια. Γιατί εμεί στη τελική ανάλυση θα υπονομεύσουμε το ίδιο το δίκαιο. Έτσι λοιπόν, με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια χειρίζεται το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ακριβείς δηλώσεις πιστές στην πραγματικότητα. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Δεν πρόκειται όμως να κάνουμε ανακριβείς δηλώσεις και παραπλανητικές για τους πολίτες ό,τι αφορά την νομική τάξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κοινή ευθύνη και νομίζω ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός ε, η διατύπωση ανακριβών δηλώσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νέμιτς. Να δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο Χάμαρμπερκ για μια σύντομη απάντηση. Ευχαριστώ. Α, δεν ξέρω, μου είπαν πριν ότι μιλάω πολύ. Πρώτα απ' όλα, προς την κυρία Ρενό, η φτώχεια είναι πράγματι πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε είναι πως η οικονομική κρίση είχε καταστροφικά αποτελέσματα στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και νομίζω πως πρέπει να ενταθεί η ανάλυση και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι όταν μιλάμε στη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει για να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένου, τους ανάπηρους, οικογένειες, ειδικά τις μονογονεϊκές από τις συνέπειες ε, της λιτότητας που επιβάλλεται στη μία χώρα μετά την άλλη. Είναι πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χαίρομαι για το ότι είναι εδώ πέρα η Ιρλανδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εκεί για το πώς σε μια συγκεκριμένη περίπτωση θα προστατεύσουμε ε, ευάλωτες ομάδες από τις αρνητικές συνέπειες ε, της λιτότητας. Για τη CIA και τη λογοδοσία, ναι, δεν έχουμε κάνει αρκετά, πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ε, το επιχείρημα κατά της περισσότερης διαφάνειας είναι πως εδώ πέρα κινδυνεύουν εμπιστευτικά στοιχεία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ CIA και Εθνικών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Αλλά πρέπει να πούμε πως ε, αυτή η εμπιστευτικότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να καλύψουν σοβαρές ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν μιλάμε λοιπόν για τεκμηριωμένα στοιχεία βασανιστήριων εκ πρώτης όψης, πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει ατιμορρησία. Όταν μιλάμε για συντονισμό μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, και του Μηχανισμού εκεί και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης η ε, πιθανές συνέπειες λοιπόν ένταξης της Ένωσης ε, στο, ε, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι μεγάλες και δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Νομίζω πως συμβολικά και πρακτικά υπάρχει δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που είχαμε εδώ πέρα. Για τις δύο παράλληλες διαδικασίες. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό έτσι, με πνεύμα συνεργασίας. Και βράχει πρόθεσμα είναι βεβαίως ε, ζήτημα νοοτροπιών και από τις δύο πλευρές να σκέφτω ένας τι κάνει ο άλλος. Νομίζω πως είχαμε κάποιες, κάποια ατυχή περιστατικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά η συζήτηση ένταξης είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα για την σύμβαση και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ναι, Πράγματι ο χάρτης όπως είπαμε συντάχθηκε 50 χρόνια μετά τη σύμβαση οπότε περιλαμβάνονται στοιχεία που δεν θεωρούνταν πρόβλημα πριν από 50 χρόνια αλλά το δικαστήριο του Στρασβούργου έχει την δυνατότητα με βάση τις αρχές της σύμβασης να κάνει, έχει μια εξελισσόμενη ερμηνεία για το τι σημαίνουν αυτές οι αρχές σήμερα. Τέλος δεν θέλω βεβαίω ε, τώρα να καταλάβω αυτό που θα πει ο δικαστή ο κύριος Τούλκενς, αλλά Ούτως ή έχουν αναφερθεί αυτά και σε αποφάσεις ε, του δικαστήριου του Στρασβούργου. Πέρυσι τον Ιούνιο είχα μια απόφαση, ε, μια υπόθεση από την Αυστρία που αφορούσε το δικαίωμα ζευγαριών του ιδίου φίλου να, να παντρευτούν. Και χρησιμοποιήθηκε αυτό ως βάση των, των συμπερασμάτων. Οπότε υπάρχει νομίζω βέβαια όφελος. Συμφωνώ επίσης με τη γενική περιγραφή τη νοοτροπία που περιέγραψε η Σάρα Λάντφορντ. Αυτή την νοοτροπία πρέπει να έχουμε. Δεν υπάρχει τομέα στην Ευρώπη που θα πρέπει να προστατεύεται από την παρακολούθηση ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να υπάρχει ίση αντιμετώπιση για να υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύστημα που προσπαθούμε να δείξουμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Χάμερμπεργκ. Κύριε Μπέγκερ, παρακαλώ να είστε σύντομος. να σας ευχαριστώ και για την απάντησή σας κύριε Νέμιτς. Ε, βλέπετε πως είχαν πάρα, πολύ, πάρα πολλές ελπίδες ε, όταν συντάχθηκε η χάρτα. Δεν μας άρεσε το άρθρο 51, αλλά είμαστε πραγματικά απογοητευμένοι από αυτά τα οποία συνέβησαν από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η απογοήτευσή μας. Σύντομα. Τώρα. Για τις παραδόσεις στη CIA. Τώρα υπάρχουν δεδομένα. Η Φιλανδία έδωσε και άλλα δεδομένα πτήσεων. Οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία. Βλέπουμε κρατούμενους στον Κουαντανάμο που πρέπει να πάνε αλλού. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε δραστηριότητα εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε γιατί δεν μπορεί να συμβεί αυτό και με άλλα σημεία. Η Κομισιόν έχει κάνει πράγματα, ναι, όντω, ε, έχει γράψει κάτι επιστολές αλλά δεν έδωσε ποτέ συνέχεια, γιατί δεν μπορούμε να επικαλυστούμε το άρθρο 7 όταν μιλάμε για την πλήρη απαγόρευση βασανιστήριων. Βασανιστήρια στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απάντηση δεν είναι επαρκής. Αυτό λέμε. Και υπάρχουν τα μέσα. Κατόπιν, για τον νόμο περί στην Ουγγαρία είναι φανταστικό παράδειγμα. Πρέπει να το αναλύσουμε. Ήταν σαφές που τι ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Τόμας Χάμερμπεργκ, ο εισηγητής ε, του ΟΗΕ, ήταν σαφής επίσης. Η Βουδαπέστη είπε θα ακούσουμε την Κομισιόν. Και η Κομισιόν μου είπε εμένα προσωπικά, ε, συγγνώμη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το χάρτη, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, οπότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα. Και τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, βρίσκουμε παραθυράκια. Κατόπιν, Σάρα, σε απάντηση ορισμένων πραγμάτων που είπατε. Σας ευχαριστώ, πράγματι έχετε υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι πρέπει να πω σε όλους τους ε, προβουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσπαθήστε να επηρεάσετε την κυβέρνησή σας. Προσπαθεί να καταστρέψει το μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι η μόνη, αλλά είναι οπωσδήποτε πιο ικανή. απάντηση σε κάποια σχόλια μικροφώνου. Ναι, η μεταρρύθμιση του δικαστηρίου, προσχώρηση στη συνθήκη, οδηγία για πρόσβαση σε δικηγόρο, βία κατά των γυναικών. Όπως σας είπα δεν είναι το μόνο κράτος. Πολλά κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή προσπαθούν και στον ΟΗΕ να παρεμποδίσουν και θέλουμε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Ωραία, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζω εκεί που σταμάτησαν οι προλαλήσαντες. Είναι σημαντικό και για μας τους, ε, βουλευτε... Ε, τους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και για σας ε, τους ευρωβουλευτές να προωθήσετε την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έτσι μπορούμε μόνο να συνδυάσουμε ε, τις προσπάθειές μας και να συνεργαστούμε για να δημιουργηθεί ένας κοινό χώρος προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Και ελπίζω αυτό να το πετύχουμε στο εγγύς μέλλον και όχι στο απότερο μέλλον, αλλά από εμά εξαρτάται. Και μάλιστα καλό θα είναι να προωθήσουμε την ένταξη και σε άλλες συμβάσεις. Πέρασαν 50 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πολλές συμβάσεις στο μεταξύ και πρωτόκολλα έχουν εγκριθεί. Γιατί να μην εντάξουμε και αυτά στην ε, νομοθετική βάση, την κανονιστική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ελπίζω να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και η συνεργασία μεταξύ των ε, κοινοβουλίων μας, ε, των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων στην νομοθετική διαδικασία είναι σημαντική και θα πρέπει να γίνεται συστηματικά να αποφύγουμε κενά, παραθυράκια και να μην δημιουργηθεί ένας ανταγωνισμός μεταξύ μας. Ένας ε, νομοθετικός ανταγωνισμός, γιατί τέτοιος ανταγωνισμός δεν θα εξυπηρετήσει ούτε την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ούτε και τη σωστή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Ελπίζω να καταφέρουμε να συνεργαστούμε και στην παρακολούθηση, γιατί και σε θέματα monitoring παρακολούθησης πρέπει να γίνουν πολλά, γιατί στη Συμβουλή τη Ευρώπη έχουμε σώματα που βοηθούν και φορεί που βοηθούν στην παρακολούθηση των συμβάσεων, της κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποφυγή βασανιστήριων κτλ. Οπότε η συμμετοχή και σε τέτοια όργανα θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε αυτό το πανευρωπαϊκό χώρο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επαναλαμβάνω, από εμά εξαρτάται να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας, τους επιτρόπους μας, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η αλλαγή. Ευχαριστούμε κύριε Λάντκριν και ευχαριστώ όλους ε, τους προσκεκλημένους σε αυτό το πάνελ του πρώτου μέρους της δημόσιας ακρόασης. Τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος και προσκαλώ το δεύτερο πάνελ και τους εμπειρογνώμονές μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας και τις παρεμβάσεις We will continue. Συνεχίζουμε λοιπόν. They, they know it. Thank you very much. Thank you. Thank you. invite Ας έρθει παρακαλώ το δεύτερο πάνελ, οι εμπειρογνώμονες μας στο δεύτερο μέρος της δημόσιας ακρόσης. We in Δυστυχώς δεν προβλέπεται διάλειμμα γιατί Έχουμε ξεπεράσει το ωράριό μας και δεν προλαβαίνουμε να <laughs> διακόψουμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Έγγιλ Λέβιτς, δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ τις συζητήσεις να τις συνεχίσετε εκτός αθούς. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν καλωσορίζω τον κύριο Έγγιλ Λέβιτς, δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ο πρώτος ομιλητής μας στο δεύτερο μέρος της δημόσιας ακρόασης. Κύριε Λέβιτς, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, καθίστε συνάδελφο. Ladies and gentlemen, uh, I thank you for the opportunity to speak. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ να μιλήσω σε αυτή την ακρόαση. Φυσικά θα σας δώσω την προσωπική μου άποψη και όχι την άποψη του δικαστήριου. Και να πω κάποια λόγια για το ρόλο του χάρτη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Καταρχήν, το πεδίο εφαρμογής του χάρτη που ήδη αναφέρθηκε από τον κύριο Νέμιτς αλλά και από άλλους συναδέλφους. Πρώτο θέμα, όσον αφορά την δικαστικότητα και το πεδίο εφαρμογή του χάρτη. Τα όρια προβλέπονται στο άρθρο 51 του ίδιου χάρτη. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα ανάμεσα στο περιεχόμενο του χάρτη και το πεδίο εφαρμογή του υπάρχει κάποια ένταση. Το περιεχόμενο του χάρτη προχωρά περισσότερο από το πεδίο εφαρμογή του. Αυτός ο χάρτης ε, περιλαμβάνει διάφορα θεμελιώδη δικαιώματα ε, γιατί ωστόσο το πεδίο εφαρμογή είναι πολύ πιο στενό. Φυσικά είναι ένα σύγχρονο έγγραφο ανθρωπίνων δικαιωμάτων βέβαια, αλλά σύμφωνα με τις συνθήκες μόνο ένα τμήμα αυτών μπορούσε να είναι τμήμα που να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ένωσης, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε κάποια σύγχυση για το ευρύτερο κοινό. Διότι το άρθρο 51 του χάρτη που περιορίζει το πεδίο εφαρμογή έχει συνταχθεί σε σχετικά περίπου, με σχετικά περίπλοκο τρόπο και ο περίπλοκος δικαστικός χαρακτήρας ε, του άρθρου δεν διευκολύνει την κατανόησή του. In short, the charter does not apply to... Εν ολίκης ο χάρτης δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις όπου διακυβεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι εγγυημένη τόσο από τα συνταγματικά συστήματα των κρατών μελών, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον χάρτη ο οποίος εφαρμόζεται από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σώματα και αφοράται κυρίως το νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν που πρέπει να είναι απόλυτα σύμμορφο με το χάρτη για να συμμορφούνται προς τις απαιτήσει του κοινοτικού νόμου και εφαρμόζεται και για τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης και στα κράτη-μέλη μόνο κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού, του ευρωπαϊκού νόμου, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Άρα μέσω της Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της δεσμεύονται να επεκτείνουν την εφαρμοσιμότητα του χάρτη όμως αυτό δεν είναι τόσο προφανές στο κοινό και επίσης δεν είναι τόσο προφανές ούτε στις δικαστικές κοινότητες των κρατών μελών. Δεν ισχύει ο χάρτης σε περιπτώσεις όπου η κοινωνική νομοθεσία δεν, ε, δεν ε, διακυβεύεται. Επίσης, εκεί όπου δεν ισχύει ο χάρτης, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι εγγυημένα σύμφωνα με τα εθνικά συνταγματικά συστήματα. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν κανόνες ε, που προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους οποίους εφαρμόζουν τα εθνικά δικαστήρια. Έχουμε για παράδειγμα τώρα μια υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με την άποψή μας, είναι σαφής παραβίαση του εθνικού συνταγματικού των εθνικών συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτά, γιατί δεν είμαστε αρμόδιοι για να κρίνουμε τα εθνικά συστήματα. Και επίσης αυτό ισχύει και για τον ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά συστήματα. Για μας η υπόθεση είναι εξαφής, αλλά τα χέρια του δικαστηρίου είναι δεμένα λόγω του άρθρου 51. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δεσμεύσεις υπό την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις τους υπό την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έτσι, ω τελικό καταφύγιο και αφού εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα σε εθνικό επίπεδο, μπορεί κανεί να έλθει ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Τώρα, τα πολλαπλά συστήματα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σημειώνουν την ανάγκη για σαφή διάκριση και περιορισμό των συστημάτων ώστε να παρεμποδιστούν οι συγκρούσεις μεταξύ τους. Το σημαίνει δηλαδή μεταξύ των Εθνικών Συνταγματικών Δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη μια πλευρά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από την άλλη. Ω προς αυτό θα πρέπει να σημειώσω ότι η λειτουργία του χάρτη δεν είναι να διευκολύνει την εναρμόνιση των συστημάτων προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Με άλλα λόγια, ο Χάρτη δεν δημιουργεί minimum standard, minimum προδιαγραφές που να γενικά να είναι εφαρμοστές, εφαρμοστέα, αυτός ο χάρτης φτιάχτηκε την, ε, με βάση τη, μια γνήσια ζήτηση για ομοιόμορφη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Για την Ένωση είναι σαφές πως η κοινοτική νομοθεσία δεν μπορεί να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα κάθε φορά με διαφορετικές απαιτήσεις και εθνικές προδιαγραφές προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η κοινοτική νομοθεσία και αυτό ισχύει παραπάνω όσον αφορά την εγκυρότητα της κοινοτική νομοθεσίας. Το να κάνουμε κάτι διαφορετικό θα δημιουργούσε τον κίνδυνο της ύπαρξης 27 διαφορετικών στάνταρ προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντό της Ένωσης. Και άρα ανομοιόμορφη εφαρμογή της κοινοτική νομοθεσίας. Είναι σημαντικό ο σεβασμό για την ομοιόμορφη εφαρμογή τη κοινοτική νομοθεσία στα κρατη Είναι ωστόσο προφανέ επίση, κατά την άποψη του δικαστηρίου, πω οι υποχρεώσει των κρατών μελών να σέβονται τι διατάξει του χάρτη απαιτούν την εφαρμογή της ε, κοινοτική νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο. Και η προηγούμενη συζήτηση επέδειξε το ίδιο πρόβλημα. Το πρόβλημα δηλαδή του χάρτη ε, που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 51 και 52. Δεν υπάρχει ο στόχος της επικάλυψης των διατάξεων των εθνικών συνταγμάτων που εφαρμόζουν το Γενικό Σύστημα Προστασίας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όπως αυτό αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι κατακλείδη ο χάρτης συμπληρώνει αλλά δεν αντικαθιστά τα εθνικά στεγματικά συστήματα, το σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτό το εγγυάται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα, εφαρμογή του χάρτη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αν και αυτός ο χάρτης έρθει να ισχύει πριν από δύο χρόνια μόλις, το, το Δικαστήριο ήδη έχει εκδώσει αρκετές αποφάσεις, 55 με 60, με παραπομπή στον χάρτη. Οι σχετικές αποφάσεις ποικίλουν. Ιδιαίτερα στα θέματα κοινωνικής πολιτικής, στα θέματα ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων, το καθεστώ των προσφύγων και ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Πολλά θέματα θα πρέπει να λυθούν με βάση την ομολογία του ΔΕΚ. Ιδιαίτερα αυτό το έργο του ΔΕΚ είναι εγγενές σε όλες τις ευρωπαϊκές διατάξεις όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων διότι αυτές οι διατάξεις διατυπώνονται με αόριστο τρόπο και άρα χρειάζεται να συγκεκριμενοποιηθούν μέσω της νομολογίας. Παραδείγματο χάρη, το δικαστήριο τώρα σε διάφορε υποθέσει, έχει να αντιμετωπίσει το κέριο ερώτημα τη πρακτικής εφαρμογής του χάρτη μέσω οριζόντια επίπτωση. Αν δηλαδή ένας ιδιώτης μπορεί να, να χρησιμοποιήσει το χάρτη, να επικαλεστεί το χάρτη απέναντι σε έναν άλλον ιδιώτη. Τον Ιανουάριο θα αποφασίσουμε για αυτό το θέμα. Αν μου δίνετε λίγο ακόμα να, εξηγήσω ακόμα κάτι. Τρία λεπτά μου δίνετε ακόμα, μάλιστα. Από όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν με το χάρτη, θα ήθελα μέσα σε τρία λεπτά να σας πω ένα παράδειγμα για το έργο του δικαστηρίου για την εφαρμογή του χάρτη, για να γίνει διάκριση ανάμεσα στις, ε, στα δικαιώματα και τις αρχές. Η διάκριση εισάγεται από το άρθρο 51, παράγραφος 1, δεύτερη φράση. Οι ηλικέ διατάξει του χάρτη, ωστόσο, δεν υποδεικνύουν αν είναι αρχές, μάλλον δικαιώματα ή αρχές. Στο άρθρο 52 λέει ότι τα υποκειμενικά δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά, ενώ οι αρχές θα πρέπει να τηρούνται. Μια πολύ λεπτή διάκριση, αλλά πολύ σημαντική διάκριση. επεξήγηση τώρα παραπέμπει στην ομολογία του ΔΕΚ καθώς και στην ομολογία των κρατών μελών και τα συνταγματικά του συστήματα. Ιδιαίτερα στο το πεδίο των κοινωνικών δικαιωμάτων και δηλώνει ότι οι αρχές δεν δίνουν ε, λαβή για άμεσες απαιτήσεις για θετική δράση από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή από τις αρχές των κρατών μελών. Άρθρο 52 Παράγραφος 5 παρέχει, τις, ε, προβλέπει μάλλον ότι οι αρχές μπορεί να εφαρμοστούν από τους θεσμούς, τους φορείς, ε, τους οργανισμούς τις Ένωσες και τα κρατημέλη όταν εφαρμόζουν το, την κοινοτική νομοθεσία στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. ότι <coughs> όλα αυτά θα είναι αναγνωρίσιμα μόνο στην ε, ερμηνεία, μόνο στην ερμηνεία τέτοιων πράξεων στην απόφαση για την νομιμότητά τους. Η διάκριση ανάμεσα στα δικαιώματα και τις αρχές θα έπρεπε να μειώνει τις αποκλήσεις ανάμεσα στις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών και να τις οδηγήσει σε ένα κοινό παρανομαστή. Και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο τη αντιφατική συζήτηση όσον αφορά τι προδιαγραφέ για υποκειμενικά δικαιώματα και αντικειμενικά δικαιώματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, των οποίων η δυνατότητα εκδίκασης έχει αμφισβητηθεί από τη σύμβαση είναι πολύ σημαντική. Η διαφορά ανάμεσα στις διάφορες θέσεις εξηγείται από τις διαφορετικές πολιτικές ευαισθησίες και τις διακεκριμένες χωριστές ε, συνταγματικές παραδόσεις όσον αφορά την ύπαρξη των υποκειμενικών και αντικειμενικών δικαιωμάτων και κυρίως των κοινωνικών δικαιωμάτων. Όπως είπα, ο χάρτης δεν χαρακτηρίζει με μονομένα άρθρο όσο ότι αυτά συστήνουν συγκεκριμένα δικαιώματα ή αρχές. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, ένα τέτοιο χαρακτηρισμό εξαρτάται από τη μελλοντική νομολογία του ΔΕΚ που θα Ε, λάβει υπόψη τις κατευθύνσεις που δίνονται στις επεξηγήσεις. Ο χαρακτηρισμός των άρθρων του χάρτη ως αρχών δικαιωμάτων ή και των δύο δεν είναι εύκολος. Το ΔΕΚ έχει να αντιμετωπίσει το θέμα του ποια στάνταρ αναλυτικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να χαρακτηρίσει το κάθε άρθρο. Δεδομένης της διατύπωσης του άρθρου 52 παράγραφος 5, οι σχετικέ επεξηγήσεις και η προέλευση της διάκρισης ανάμεσα στις δικαιώματα και αρχές αυτό το χάρτη, είναι σαφές ότι δεν συνιστούν υποκειμενικό δικαίωμα το οποίο να μπορούν να επικληθούν άτομα. Η Πρόεδρο ζητεί να συντομεύσετε. Όσον αφορά τι επιπτώσει για την δικαστική αναθεώρηση για την παραβίαση δικαιωμάτων και αρχών, το γεγονό ότι οι προ, διατάξεις δεν συστήνουν ε, ε, δικαιώματα, μπορούμε να πούμε ότι είναι και περιορισμένη η δυνατότητα επίκλησής του στο δικαστήριο. Αν χρειάζεστε τώρα επεξηγήσεις μπορώ να σας ε, τις δώσω αργότερα. Σας ευχαριστώ δικαστή Λεβίτση, και ελπίζω ότι στη συζήτηση θα μας διευκρινίσετε τις απορίες μας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο Ολκίνης, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση γιατί μας επιτρέπει να συνεχίσουμε στι Βρυξέλλες τον πολύ καρποφόρο διάλογο που ξεκινήσαμε στο Στρασβούργο μεταξύ της Επιτροπής σα και της Ευρω... του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, γιατί σίγουρα σε θέματα δικαιωμάτων και ελευθεριών έχουμε ε, κοινό ενδιαφέρον. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, είναι ένα εργαλείο με διπλή και μεγάλη σημασία. Καταρχήν, σε συμβολικό επίπεδο, ο χάρτης έχει διατρανώσει την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εδράσει την εξουσία και να εντάξει την δράση της στην νομιμότητα που χορηγεί αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και σε πρακτικό επίπεδο, ο χάρτης δεσμεύει την Ένωση να αναλάβει δράση, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά, να προστατεύσει, σεβαστεί, να αναπτύξει και να πραγματοποιήσει, δηλαδή και στα αγγλικά του respect, protect, promote and fulfill, τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα. Έτσι δίνει την έμφαση στις υποχρεώσεις της Ένωσης που μπορούν ίσως να δημιουργήσουν μια διαγραφή των διαφόρων όριων μεταξύ πολιτικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι και το σημαντικό ενδιαφέρον του χάρτη. Φυσικά υπάρχει υποχρέωση σταδιακής εφαρμογής και υλοποίησης του χάρτη, οπότε το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε όλες τις προσπάθειες που θα μπορούσαμε να πετύσουμε από αυτή, στα πλαίσια φυσικά των αρμοδιοτήτων της ε, για το χάρτη και το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 51 που ακούσαμε στη διάρκεια της ακρόασης. Στα πλαίσια της διαμόρφωσης μιας Ευρώπης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε τι φάση βρισκόμαστε. Κατά τη γνώμη και από το πρίσμα μάλλον της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και απόψη δικαστηρίου που πρέπει να εξασφαλίσει το σεβασμό αυτής, αυτού του αυτή τη ευρωπαϊκή σύμβαση θα ήθελα να πω το εξή ό,τι αφορά την συνύπαρξη του χάρτη και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ε, θα μιλήσω στη συνέχεια για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο οργάνων και τέλο για το συμπλήρωμα της συμπληρωματικότητα και συγχωρήστε με για το λογοπαίγνιο. Καταρχήν θα πρέπει να, ε, να λάβουμε υπόψη ότι τις εργασίες του χάρτη που έγιναν μεταξύ 1999 και 2000 και να δούμε πώς διαμορφώνονται σήμερα με τις ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ των ε, πολιτικών δυνάμεων και παρακολουθήσαμε με ζωντανό ενδιαφέρον αυτή τη συμφωνία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το 1999 2000 η συνύπαρξη χάρτης και ε, χάρτας και Ευρωπαϊκής Σύμβασης δημιούργησε κάποιες επιφυλάξεις. Στο πρίμιό της ε, ο χάρτης λέει ότι επανεπιβεβαιώνει τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πολιτικών Ελευθεριών και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και μια και μιλάμε για αστικά και πολιτικά δικαιώματα, αυτά τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο χάρτη, σε, στη μεγαλύτερη περίπτωση αναφέρονται ως δικαιώματα που μπορεί να καλεστεί στο δικαστήριο, αλλά τα περισσότερα ε, απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και βλέπουμε εδώ ότι οι εργασίε των συντακτών της, ε, του χάρτη δείχνουν την τεράστια δυσκολία που προϋπέθεται η διεύρυνση του καταλόγου των δικαιωμάτων που μπορεί κανείς να επικαλεστεί στο δικαστήριο και μάλιστα σε μια ένωση που τότε απαρτίζονταν από 15 χώρες. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ε, υιοθετήσει το σκληρό πυρήνα των δικαιωμάτων αυτών που κατοχυρώνται σήμερα στο χάρτη, αν προηγουμένως δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και τη συναφή νομοθεσία. Γιατί πιστεύω ότι και τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, τα βήματα είναι σταδιακά. Καταρχήν, ε, στο μεταξύ είχαμε διάφορες ε, αλλαγές και είχαμε και απλουστεύσεις και συμπληρώσεις. Γιατί είναι σημαντικό στην τρίτη χιλιετία να έχουμε καλύτερη ε, κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί οι αποδέκτες τους δεν είναι μόνο οι νομομαθείς. Γι' αυτό και στην ε, σύμβαση ε, και στο, στο χάρτη μάλιστα έχουμε όλες τις, τους περιορισμούς, τις απαριθμίσεις, λέμε το άρθρο 6, δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το άρθρο 5, δικαίωμα σε ελευθερία και ασφάλεια και φυσικά τα θέματα οικογένειας, θρησκείας, δικαιώματος εταιρείστη κλπ. Ο χάρτης λοιπόν έχει σημαντική ε, ε, λειτουργία την παραμπομπή στον στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση γιατί ο χάρτης σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εξασφαλίζει ε, ίσον προστασία από ότι η Σύμβαση. Φυσικά ο χάρτης διευρύνει το, το πεδίο εφαρμογή του, της Σύμβασης, άρθρο 14, το δικαίωμα στην παιδεία, ένα νέο ε, δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, η πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και τη δυνατότητα ε, δωρεάν παρακολούθησης της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Και είναι πολύ θετικές αυτές οι αλλαγές που απορρέουν είτε από, την, από το κοινοτικό δίκαιο ή από την κοινοτική νομολογία. Επίσης, ε, περιλαμβάνονται κάποια δικαιώματα στο χάρτη που δεν είχαν αναγνωριστεί ως δικαιώματα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αλλά έχουν αναγνωριστεί από την ομολογία. Γιατί η νομολογία ερμηνεύει τα κείμενα. Δεν μπορεί να είναι η σύμβαση ε, σαν ε, χειρόγραφο της νεκράς θάλασσας. Επίσης έχουμε το δικαίωμα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστη, αυτά τα νέα δικαιώματα. Η απαγόρευση, και αυτό είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου, απέλασης σε ε, χώρα που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποστεί κακή μεταχείριση. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δικαιώματα. Από όλα αυτά τι προκύπτει. Έχουμε δικαιώματα που στο χάρτη προσφέρουν ε, και κατοχυρώνουν ε, άλλες φορές μεγαλύτερη προστασία και άλλες φορές κατώτερη προστασία από αυτή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Βέβαια αυτό συνάδει με το άρθρο 53 της Σύμβασης που λέει ότι η Σύμβαση είναι το ελάχιστο και ζητούμε από τα υπόλοιπα όργανα να ενισχύσουν αυτό το ελάχιστο, την ελάχιστη προστασία. Βέβαια, αυτό που επίση είναι σημαντικό και το αναφέρατε και εσεί πριν από λίγο, είναι ότι σε πολλές αποφάσεις του δικαστηρίου, όλο και περισσότερο, όταν βλέπουμε στο χάρτη πιθανότητα ενίσχυση του επίπεδου προστασίας, φυσικά και θα το κάνουμε. Έγινε αυτό στην περίπτωση των φιλομεταβατικών ή το θέμα της αναδρομικότητας των θετικών ποινικών δικαιωμάτων ε, ή σε θέματα γάμου. Όταν υπάρχει δυνατότητα μέσω του χάρτη να ενισχύσουμε την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το κάνουμε. Και μάλιστα ο χάρτης έχει και, δίνει και ναύσματα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Και υπάρχει μια αμοιβαία τροφοδοσία μεταξύ των δύο ε, νομοθετημάτων. Βέβαια, θα πρέπει να αποφύγουμε τη δεύτερη περίπτωση, η ίσονο προστασία. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο και πολιτικά, αλλά και νομικά συμβίβαστο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Γι' αυτό έχουμε και την περίφημη Γενική Διάταξη του Χάρτη. Η Γενική Διάταξη του άρθρου 52 παράγραφος 3 λέει ότι στο μέτρο που ο χάρτης περιλαμβάνει αντίστοιχα δικαιώματα με αυτά της Σύμβασης, το νόημα και η εμβέλεια των δικαιωμάτων αυτών είναι παρόμοια με αυτά της σύμβασης. Πολύ σημαντική αυτή η διάταξη. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν αποδέχεται ασθενέστερη προστασία του χάρτη. Και μάλιστα έτσι εξασφαλίζεται η συνάφεια μεταξύ χάρτη και Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και όλες αυτές οι εξηγήσει αναφέρονται και στη σύμβαση αλλά και στα πρωτοκολλά της αλλά και περιλαμ... καλύπτουν και την ομολογία. Συνοψίζω λοιπόν, ο συντάκτης ε, του χάρτη ενέταξε το χάρτη σε μια συνέχεια ως προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δεύτερον, συμπληρωματικότητα μεταξύ χάρτη και Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ε, το ΔΕΚ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακόμη και πριν γίνει υποχρεωτική αυτή η συμπληρωματικότητα, εμείς την εφαρμόζαμε. Και μάλιστα ο πρόεδρος Κουρίς ε, του, ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ο κύριος ε, Κώστα έχουν συντάξει από κοινού ένα έγγραφο και μία, σε μια κοινή επιτροπή στην οποία είπαν ότι θα έπρεπε να μεριμνήσουμε για να εξασφαλιστεί συνάφεια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και του Χάρτη. Και στα πλαίσια αυτού του άρθρου 52 παράγραφος 3 που σας ε, διάβασα πριν από λίγο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια παράλληλη ερμηνεία των δύο κειμένων που κρίνεται απαραίτητη. Από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, τότε που βλέπουμε, παρατηρούμε και τις πρώτες εφαρμογές του άρθρου 52 παράγραφος 3 του χάρτη, ακριβώς αυτό το, την κατεύθυνση ακολουθούμε. Ε, ο Άγγιλ ε, Λεβί ήταν προηγουμένω ε, και δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν ξέρω αν συμφωνεί. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική αυτή η κατεύθυνση. Καταρχήν, κάποιε εφαρμογέ. Έχουμε την τη... Τη... μια απόφαση του 2000, 5 Οκτωβρίου 2010, για τη συνεργασία σε θέματα αστικού δικαίου και κυρίω την ερμηνεία του της έννοιας του δικαιώματος δαιμονία των παιδιών σε περίπτωση που δεν είναι τα παντρεμένοι γονείς. Η σύμβαση λέει, όπως προκύπτει το άρθρο 52 παράγραφος 3, σε περίπτωση που έχουμε αντίστοιχα δικαιώματα με αυτά που κατοχυρώνονται στην σύμβαση, το νόημα και η εμβέλειά τους είναι η ίδια. Βέβαια, η, η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει το κοινοτικό δίκαιο να χορηγήσει ακόμη πιο ενισχυμένη προστασία. Βέβαια, όταν εξετάζουμε την ομολογία αυτή και το δικαίωμα των ε, δικαστών, είναι σημαντικό να δούμε τα επιπλέον στοιχεία. Μία άλλη απόφαση του 2010 μιλάει για την προστασία των φυσικών προσώπων σε ό,τι αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Είναι θέμα ιδιωτικού βίου. Και πάλι το δικαστήριο είπε ότι εφαρμόζεται το άρθρο 52 παράγραφος 3 και το άρθρο 53 των Γενικών Διατάξεων που λένε ότι καμία διάταξη του χάρτη δεν μπορεί ή δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως περιοριστική των ε, δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Σε μία άλλη απόφαση κατά της Γερμανίας για την ε, προστασία, την πραγματική προστασία των δικαιωμάτων της Ένωσης και κυρίως το δικαίωμα σε πρόσβαση σε δικαστήριο και σε δικαστική αρρωγή και για πρόσωπα φυσικού και ε, για φυσικά και για νομικά πρόσωπα και εκεί λαμβάνεται υπόψη η νομολογία του ΔΕΚ. Δεν πρόκειται να σας διαβάσω όλες τις αποφάσεις. Είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου. Εκεί αναφέρεται το θέμα της ε, ε, α, μεταφοράς των ετούντων άσυλων στο κράτος υποδοχής, το πρώτο κράτος υποδοχής είχαμε, ε, είχαμε υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και προδικαστικό ζήτημα. Είχαμε το, την περίπτωση Ελλάδας-Βελγίου MSS ε, που το δικαστήριο έκρινε ότι η επαναφορά ε, σε χώρα που υπήρχε κίνδυνος για κακή μεταχείριση δεν επιτρέπεται. Και αυτό που βλέπουμε στην απόφαση NS του Λουξεμβούργου, βλέπουμε τα συμπεράσματα του Γενικού Εισαγγελέω που ακριβώ έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Σε ό,τι αφορά το μεθοδολογικό επίπεδο, έχουμε φυσικά τι βασικέ αρχέ, τι γενικέ αρχέ. Παρακαλώ, έχετε ξεπεράσει το χώρο σας. Λέμε απλώς ότι ε, η ερμηνεία θα πρέπει να είναι δυναμική γιατί και η νομολογία είναι δυναμική και ως προς την ουσία της η απόφαση στα συμπεράσματα του Γενικού Σαγγελέως μιλάει ότι χρειάζεται συμπληρωματικότητα με την προηγούμενη απόφαση MSS. Τρίτο σημείο, συμπλήρωμα της συμπληρωματικότητας. Αυτή είναι, αυτό είναι η ένταξη τη Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Στην αρχή υπήρχε μεγάλη απεσιοδοξία, αλλά τελικά συνέβη το αντίθετο. Θεωρούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή ε, σύμβαση θα ήταν το αντίθετο και τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι το αντίθετο, απλώ είναι το λογικό συμπλήρωμα του χάρτη και η συνθήκη της Λισαβόνας είναι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένταξη προσχωρεί στη σύμβαση, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα υπάρχουν κάποια κείμενα που εξετάζονται και πολύ σωστά κυρία μου είπατε πριν από λίγο ότι υπάρχει πολιτική βούληση για την ένταξη ήδη από τη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά οι πρακτικοί τρόποι υλοποίησή τη ακόμη συζητώνται. Θα πρέπει πάντως να φέρουμε και πάλι επιτάπητο στο θέμα και να ανανεώσουμε την πολιτική βούληση της ένταξης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί έτσι μόνο θα δημορφωθεί ένας πραγματικά δημοκρατικός χώρος προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη αν υπερεύει το ωράριό μου. Σας ευχαριστούμε κυρία Τάλκενς. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Περνάμε αμέσως στον επόμενο ομιλητή, ο οποίος εκπροσωπεί την υπηρεσία για τα... τον Οργανισμό για Θεμελία Δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Γκαμπριέλ που Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Να ξεκινήσω ναι, συγχαρητήρια. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ ε, σημαντική αυτή η συζήτηση και η πολιτική όθηση που χρειάζεται κάθε χρόνο και δεν βλέπω εγώ κάποια αλληλεπικάλυψη μεταξύ των εκθέσεων που έχουμε κάθε έτος. Έχουμε την έκθεση της Κομισιόν, της υπηρεσίας μας και την έκθεση του Κοινοβουλίου. Και θεωρώ πως η σχέση μεταξύ αυτών των τριών εκθέσεων είναι μια συμβιωτική σχέση. Θα έλεγα πως ε, η μία γονιμοποιεί την άλλη και όπως βλέπετε στην τελευταία μας έκθεση προσθέσαμε ένα νέο κεφάλαιο το υπαρτιμό 10 που αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και αυτό έγινε με βάση το δικό σας ψήφισμα και αναφέρθηκε ήδη το θέμα αυτό π.χ. ο κύριος Λέβιτς ο δικαστής είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πλήρη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου της Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Τον κύριο Σχαμαρμπεργ και η κυρία Λούντ μιλούσαν για προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συνεργασία Συμβουλίου της Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να κάνω είναι να σας παρουσιάσω τα νέα δεδομένα μας για τη νέα έκθεση του 2011. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τα δεδομένα ήταν πριν από δύο ημέρες στη βγαίνει και τα επεξεργαζόμαστε, αλλά δεν θα πρέπει βεβαίως να σας απογοητεύει αυτό, καθώς όπως ξέρετε το 2011 δώσαμε πάρα πολλά δεδομένα και αναλύσεις στο Κοινοβούλιο που αντιμετωπίζουν τις βασικές προκλήσεις που θεωρήσαμε σημαντικές. Θα αναφέρω γρήγορα και γρήγορα 7 από αυτές. Πριν από μία εβδομάδα ένας συνάδελφός μου παρουσίασε στην Επιτροπή σας μία έκθεση για την κατάσταση παρατύπων μεταναστών και τα νομικά και, προβλήματα, και άλλα προβλήματα που είχαν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ε, είχαν συζητηθεί και εδώ πέρα αυτά τα ζητήματα. Πολιτική συμμετοχή ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και διανοητικής ε, αναπηρίας και εδώ πέρα υπάρχουν πολλές ε, προκλήσεις ε, το 2011. Τον Ιούνιο δε είχα ξαναέρθει εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο και παρουσίασα την έκθεσή μας που εξετάζει την δυνατότητα των ε, μειονότητες από την συνθήκη της Λισαβόνας κατόπιν ετήματος του Κοινοβουλίου και εδώ πέρα είδαμε προκλήσεις αλλά και θετικές δυνατότητες. Επίσης παρουσιάσαμε βρήματα για την κατάσταση στα ελληνικά χερσαία σύνορα θα επίσης ε, ζητήματα στην αγορά εργασίας, ε, διακρίσεις στην αγορά εργασίας, αλλά εστιάσαμε και σε ένα ζήτημα που είναι σημαντικό για όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, που νομίζω άρα ταιριάζει με το πάνελ σας. Τα ευρήματα λοιπόν ήταν πως ναι πράγματι μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας η πρόσβαση στη δικαιοσύνη βελτιώθηκε στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά ακόμα υπάρχουν πολλές ελλείψεις στο επίπεδο των κρατών μελών ε, με κυριότερο το ότι είναι πολύ μακροσκελείς οι διαδικασίες ε, και δεν είναι μόνο η συνήθιση υπόπτη, είναι γενικότερο το ζήτημα. Επίσης το υψηλό κόστος για δικηγόρους και τα δικαστικά έξοδα ένα άλλο ζήτημα και βεβαίως περιοριστικοί κανόνες για το ποιος μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Συνοψίζοντας, νομίζω πως το 2011 έχουμε αποστείλει πολλά στοιχεία στο Κοινοβούλιο από την υπηρεσία μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως στην τελευταία έκθεση ζητήσατε από τα θεσμικά όργανα που λαμβάνουν τις αποφάσεις να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά. Θυμάμαι πως δώσαμε και δύο γνωμοδοτήσεις. Το Κοινοβούλιο μία φορούσε την οδηγία για τα δεδομένα αεροπορικών επιβατών και άλλη μία για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα έρευνη. Ελπίζουμε να ήταν χρήσιμο και για να τελειώσω, είδατε, είδατε πόσο γρήγορο είμαι, να τονίσω πως δεν είναι σημαντικό μόνο να περιγράφουμε την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά ίσως είναι πιο σημαντικό να κοιτάμε και τις τάσεις που υπάρχουν στην εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε κάποιους δείκτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δικτών είναι το πλαίσιο της ε, Κομισιόν για τις Εθνικές Στρατηγικές Εσωμάτωσης των Ρωμά που αναφέρθηκαν ήδη εδώ πέρα η Κομισιόν ζήτησε από την υπηρεσία μας να επεκτείνει την ερευνά της και να παρακολουθήσει τα επόμενα 8 χρόνια την πρόοδο επιτόπου. Και τελευταία μου παρατήρηση, εδώ πέρα μπορούμε, μπορεί η υπηρεσία μας να προσφέρει μια προσθέμενη αξία γιατί δεν ε, εξετάζουμε τόσο πολύ την αξιολόγηση, την νομική συμπεριφορά των κρατών μελών αλλά την κατάσταση των ανθρώπων. Δηλαδή ένας κλασικός φορέας ε, θα εξέταζε ε, τα κρατη και τη, αυτούς που είναι υποχρεωμένοι δηλαδή να διαφυλάξουν τα δικαιώματα. θα κοιτάμε του φορεί των δικαιωμάτων, δηλαδή των ανθρώπων. Ανέφερα ήδη τις γυναίκες ΛΟΑΤ, ε, του Εβραίου και όσον αφορά την βία για τις γυναίκες θα πάρουμε συνεντεύξεις από 40.000 γυναίκες για τις εμπειρίε τους και νομίζω πως πάλι αυτά τα δεδομένα μπορούν να σας βοηθήσουν στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήσασταν γρήγορος και περνάμε αμέσω στον κύριο Έμον Μακαόντα επικεφαλής της Ιρλανδικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι γρήγορος. Νομίζω πως είναι η δεύτερη φορά τον τελευταίο 1,5 χρόνο που έχετε προσκαλέσει εθνικά θεσμικά όργανα και χαιρόμαστε για το ότι είμαστε και πάλι σήμερα εδώ πέρα. Πέντε πράγματα θα ήθελα να πω τα επόμενα λεπτά. Να μιλήσω λίγα για τα θεσμικά όργανα ανθρώπινων δικαιωμάτων κατόπιν ε, για την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εθνικών ε, Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ήμασταν μέχρι πριν από λίγους μήνες πρόεδρος, τώρα είναι η Σκοτσέζικη Αρμόδια Επιτροπή. Κατόπιν θα δούμε τη σημασία του χάρτη για τη δουλειά μας. Τέταρτον, να δούμε τις συστάσεις των Ευρωπαϊκών Ομάδων και τις προτεραιότητες μας. Τώρα για τα εθνικές αυτές υπηρεσίε. Οι αρμοδιότητες μας ε, περιλαμβάνουν νομοθετική έρευνα, έρευνα, χάραξη πολιτικής, εκπαίδευση, κατάρτιση, νομικές παρεμβάσεις, οπότε είναι αρκετοί οι φορείς. Είναι φορείς ε, με μια νομική συνταγματική βάση που βασίζεται σε αρχές του ΟΗΕ για να έχουν μια ευρεία εντολή και να είναι ανεξάρτητη. Οπότε είμαστε κάτι τρίτο μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και κράτους. Χρηματοδοτούμαστε από το κράτος, αλλά είμαστε ανεξάρτητοι από αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει 36 μέλη από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 22 έχουν το λεγόμενο καθεστώ Α, δηλαδή συμμορφώνονται πλήρω με τις αρχές του ΟΗΕ. Εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 18 τέτοιες, ε, τέτοιοι φορεί. Μπορεί να είναι μια επιτροπή, συνήγορος. Το βασικό είναι να είναι ανεξάρτητο. ο φορέα. Έχουν λοιπόν διαφορετικές έντολες, αλλά όλες έχουν το λεγόμενο καθεστώς Α, σύμφωνα με τις αρχές των Παρισίων, έχουν την δυνατότητα να σχολιάζουν ε, νομοσχέδια. Αυτό είναι βασικό. Αυτό σε γενικές γραμμές. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ομάδα, πρόκειται για μια περιφερειακή βεβαίως ομαδοποίηση και εκεί πέρα είμαστε σε τακτική επαφή με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΗΕ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία και ως παράδειγμα του τι δουλειά κάνουν ε, οι φορείς αυτοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεργαζόμαστε π.χ. Για, τα, για τους μετανάστες, για τα δικαιώματα ΛΟΑΤ, για κακομεταχείριση αστυνομία, ε, κακομεταχείριση παιδιών, ευπαθή άτομα, σωματεμπορία κτλ. Όσον αφορά το χάρτη και τη σημασία του για εμάς. Μέχρι στιγμής ήταν περιορισμένη. Νομίζω πως αυτό οφείλεται στο ότι το πεδίο εφαρμογή ε, του χάρτη ακόμα δεν είναι σαφές ε, στα κράτη-μέλη. Επίσης, πολλά από τα δικαιώματα που καλύπτονται από το χάρτη βεβαίως καλύπτονται ε, και με εσωτερική νομοθεσία. Ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος. Συγκεκριμένη δουλειά που κάνουν τώρα πολλοί τέτοιοι φορείς σε φυλακές, η σχέση με τα παιδιά δεν συνδέεται ίσως έτσι άμεσα με το χάρτη και όπως είπαν ήδη και οι προλαλήσαντες, η ερμηνεία του χάρτη συνεχίζει ακόμα να μην υπάρχει. Είχαμε σημαντικές περιπτώσεις όπως η υπόψη Ζαμπράνο ε, για τη μετανάστευση και νομίζω πως είναι το χρόνο ο χάρτης θα ε, αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία και στα κράτη-μέλη. Τώρα η ευρωπαϊκή ομάδα μας όσον αφορά τις συστάσεις μας θα ήθελε να προωθήσει την ε, αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών. Το δεύτερο το οποίο θα θέλαμε θα είναι να ενημερώσουμε περισσότερο για τον χάρτη ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επίσης σημαντική θα είναι τεχνική αρρωγή από την Κομισιόν και οι όπω όπως σημερινή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικές για να αυξηθεί η ενημέρωση ε, στους εθνικούς φορείς σε σχέση με το χάρτη και το σημαντικό ρόλο που παίζουν ε, για την μετακένωση, αν θέλετε, στο εθνικό πλαίσιο του χάρτη. Υπάρχουν και άλλες συστάσεις, δεν θα τις αναφέρω, νομίζω πως ε, Αυτέ οι τέσσερι είναι σημαντικέ. Όσον αφορά τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκής Ομάδας ε, Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ελπίζουμε να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ε, συμμετοχής μας ως παρατηρητές στι ενταξιακέ διαπραγματεύσει ε, όσον αφορά την ΕΣΔΑ και θα απευθύνουμε επιστολή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, όσον αφορά τον ρυθμό της ένταξης. Κάτι άλλο επίσης, στο οποίο φιλοδοξούμε να δραστηριοποιηθούμε, είναι η παρακολούθηση της ε, Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Άλλο κάτι το οποίο είχε αμεθύξει ο Ιρλανδικός φορέας είναι η εξέταση της νομοθεσίας από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από νωρίς ήδη και τέταρτο και τελευταίο για εμάς θα είναι μια παρέμβαση ως αμήκους κουριεφίλη του δικαστηρίου αφού κυρωθεί από την Ένωση η σύμβαση βεβαίως. Νομίζω λοιπόν ήμουν Σύντομο και παρουσίασα κάποιες ιδέες στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μακάοντα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σύντομο. Τώρα θα ζητήσω από την Judith Sutherland, ερευνήτρια του Human Rights Watch, να αναλάβει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας και θα ήθελα να σχολιάσω και κάποια από τα όσα ακούσαμε στην πρώτη, στο πρώτο πάνελ. Όπως γνωρίζετε υπήρξε μια μεγάλη περίοδος αισιοδοξία με τη συνθήκη της Λισαβόνας και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και με την δημιουργία του χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και επίση μιλήσαμε για πολιτική μηδενική ανοχή για τα... έγινε μάλλον για πολιτική μηδενικής ανοχής για τα κράτη τα οποία παραβίαζαν αυτό το χάρτη. Δυστυχώς με τον καιρό αποδυναμώθηκε ο χάρτης και μειώθηκε και η αισιοδοξία. Τονίστηκαν περισσότερο οι περιορισμοί παρά τα θετικά στοιχεία του χάρτη. Η Επίτροπος Ρέντινγκ τόνισε τότε που εκδόθηκε η σχετική έκδοση ότι ο χάρτης αυτός ήταν περισσότερο μια πηξίδα και όχι ε, κάτι το υποχρεωτικό. Επίσης η κατάσταση των Ρώμα είναι κάτι που αποδεικνύει τα όσα λέγατε. Όπως γνωρίζετε η Επίτροπος Ρέντινγκ ε, κράτησε πολύ στεναρή στάση μέσα στην ε, μεγάλη δημοσιότητα εκστρατεία για απέλαση των Ρωμά από τη Γαλλία στη Ρωμανία κυρίως, αλλά και στη Βουλγαρία. Τότε η Ρέντινγκ ε, αντέδρασε πολύ έντονα μέσω μιας διοικητικής εγκυκλίου που δόθηκε στον τύπο, εγκύκλιο από, που εκδόθηκε στις 5 Αυγούστου από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι οι νομάρχες θα έπρεπε να λάβουν δράση ώστε να απελάσουν άμεσα όσους παρανόμως διέμεναν στη γαλλική επικράτεια και να τους δώσουν ε, να τους απελάσουν άμεσα. Θα πρέπει να είναι γνωστό ότι η απέλαση των Ρωμά από τη Γαλλία χωρίς τις ε, κατάλληλες ε, δικλείδες ασφαλείας δεν ξεκίνησε το 2010. Αντίθετα, η ΜΚΟ ήδη είχαν έρθει σε επαφή με την Κομισιόν από το 2008 με επίσημη καταγγελία αλλά δεν είχε ποτέ γίνει κάτι σε σχέση με αυτή την καταγγελία. Το νέο στοιχείο ήταν η μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε σε αυτή την εκστρατεία και ο πολιτικός χαρακτήρας που δόθηκε στην όλη υπόθεση που ήταν πολύ ανησυχητικός. Ε, αυτή τη φορά λοιπόν αντέδρασε η Κομισιόν και απείλησε τη Γαλλία με διαδικασία επιπαραβίαση των συνθήκων και ζήτησε εξηγήσει για το κατά πόσο αυτό ήταν συμβατό με την οδηγία περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Η Γαλλία επιλεκτικά είχε μεταγράψει την σχετική οδηγία. Εισήχθησαν τροπολογίες στο περί, στο νομοσχέδιο περί ε, ασύλου ε, και επίσης τον Ιούνιο του 2011 πια υιοθετήθηκε η σχετική νομοθεσία. Παρά τα μεγάλα προβλήματα αυτής της νομοθεσίας που θα σας τα περιγράψω και αποδείξεις για συνεχιζόμενες διακρίσεις κατά τον Ρωμά, από τις γαλλικές αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα, μια δήλωση φέτος τον Αύγουστο εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τα βήματα που είχε κάνει η γαλλική κυβέρνηση. Λεπτομερής ανάλυση δεν ζητήθηκε από ε, τις γαλλικές αρχές για τη σχετική νομοθεσία. Αν υπήρχε κάποιο πιο συνολικό κείμενο από ότι η δήλωση των ανακοινωθέν τύπου και μας είπαν ότι δεν χάσαμε και τίποτα. Ε, εμείς δεν συμμεριζόμαστε την εκτίμηση, της, την αξιολόγηση της Κομισιόν ούτε από νομικής άποψη ούτε στην πράξη. Έχω ένα σωρό λεπτομέρειες για την ε, νομοθεσία, αλλά νομίζω πως ε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο και μπορεί να σας κουρώσω. Γι' αυτό ίσω να μην μπω σε πολλές λεπτομέρειες και να πω απλά ότι ανησυχούμε πάρα πολύ για ορισμένε διατάξεις της νομοθεσίας που από ό,τι φαίνεται στοχεύουν τους Ρωμά για να διευκολύνουν την απομάκρυνσή του. Και αυτό συνδέεται με ένα μεγάλο αριθμό πολιτικών δηλώσεων γύρω από αυτή την νομοθεσία που σαφώς αναφέρονται στους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους, την κατάσταση στα στρατόπεδα, συγκέντρωση στον Ρωμά, τις κατασκηνώσεις μάλλον αυτών, ε, καθώς και το ε, πώς αυτά, αυτές οι κατασκηνώσεις θα χρησιμοποιούνται και από Ρωμά από άλλες χώρες της Ένωσης. Θα πρέπει να γίνουν λοιπόν μεμονωμένες αξιολογήσεις πριν ε, δίνεται η διαταγή για να απέλαση. Οι δράσεις, οι ενέργειες της Κομισιόν σε ανταπόκριση στην γαλλική κατάσταση συνοδεύεται και από την ανταπόκρισή του στη ε, κρίση δικαιωμάτων στην Ουγγαρία που συζητήθηκε νωρίτερα καθώς και στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση λοιπόν της Κομισιόν σε αυτά τα θέματα δείχνει την απροθυμία να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία επιβολής που έχει στη διάθεσή της. Έχει αναφερθεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να επενεθεί γιατί έδρασε στην Ουγγαρία από τη στιγμή που εγκρίθηκε αυτός ο πολύ προβληματικός νόμος περί ΜΜΕ εκεί ε, που λύθηκε με διαδικασίες κατά παράβαση αν με τις τροπολογίες δεν γίνονταν όλες οι απαραίτητες αλλαγές. Ωστόσο, οι αλλαγές που έγιναν το Μάρτιο άφησαν αυτό τα πιο σημαντικά προβλήματα όπως τις ευρύτατες περιορισμούς, τους περιορισμούς για τις ε, αναφορές καθώς και τις ρυθμιστικές ε, αξουσίες στα ε, κυβερνητικά ή διοριζόμενα από την κυβέρνηση σώματα και φορείς. Η Κομισιόν είπε ότι θα παρακολουθήσει την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και όπως σας είπα και το, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέο ψήφισμα τον Μάρτιο καταγγέλλοντας το ότι η Ουγγαρία δεν είχε προχωρήσει αρκετά. Επίσης, αντιμετωπίζοντας μια βαθιά κρίση μετανάστευσης και ασύλου στην Ελλάδα, η Κομισιόν δεν κατάφερε να καταλήξει κάπου, ενώ ξεκίνησε διαδικασία κατά της Ελλάδας σε σχέση με τη δυσλειτουργικό σύστημα ασύλου, καθώς και τις ε, καταχρηστικές συνθήκες ε, κράτησης των ετούντων άσυλο, η Κομισιόν τελικά δεν μπόρεσε να συνεχίσει στεναρά αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις υποθέσεις και περιορίστηκε μόνο σε τεχνική βοήθεια. Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι κάτι το συστηματικό. Και βλέπουμε λοιπόν δυσπροθυμία και διστακτικότητα να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά η Κομισιόν, που δεν διαπιστώνουμε να ισχύει η ίδια δυσπιστία σε άλλα θέματα εμπορικά ή οικονομικά, όπου η Κομισιόν επανελειμμένως και εντατικά κατηγορεί τα κράτη επί παραβάσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα πρέπει να κάνει το ίδιο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταφεύγει στη διαδικασία επί παραβάση όταν αυτό χρειάζεται. Πιστεύουμε ότι όταν υπάρχουν καταγγελίες για σοβαρή παράβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει η Κομισιόν να προβαίνει σε σοβαρά βήματα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει δώσει συμβουλές στη χώρα στην νομοθετική διαδικασία, σχολιάζοντας τα προτινόμενα μέτρα όσον αφορά την απομάκρυνση Ευρωπαίων πολιτών, ενώ θα γινόταν και κοινοβουλευτικός έλεγχος της νομοθεσίας. Και αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει κάθε φορά που η η κοινωνία των πολιτών ευρύτερα θίγουν θέμα ε, παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν να παίξουν βασικό ρόλο. Το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να ενισχύσει την ομάδα εργασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα των ανθρώπων και την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, το ΦΡΕΜΠ, e ώστε να είναι ένα αποτελεσματικό φόρουμ για την ανάλυση των προβλημάτων σε κάθε κράτος μέλος. Έχει το αντίστοιχό του όπου συζητείται η πολιτική, πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εξωτερική, στις εξωτερικές σχέσεις, την COHOM, που κάνει, έχει μια ευρεία εντολή για να συζητά την κατάσταση σε συγκεκριμένες ε, χώρες, καθώς και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες χώρες. Πιστεύουμε πως ήταν πάρα πολύ χρήσιμο η ΦΡΕΜΠ e να ενισχυθεί, να τη δοθεί σαφής εντολή, ώστε να αποτελέσει ένα φόρουμ για ανάλυση συγκεκριμένων καταστάσεων και χωρών εντός της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο πιέζει την Κομισιόν για να δημιουργηθεί η θέση του Επιτρόπου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα πρέπει να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές του, να ασκήσει πίεση στο Συμβούλιο και στα μεμονωμένα κράτη-μέλη για να στηρίξουν μια ενισχυμένη ΦΡΕΜΠ και να βοηθήσει και την Κομισιόν να ασκήσει το ρόλο της ως θεματοφύλακα των ε, συνθήκων. Μια άλλη σύσταση θα ήταν το Κοινοβούλιο να στηρίξει τη δημιουργία ενός ε, μιας θεσμοθετημένης μορφής ε, συζήτησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτή η ακρόαση, ας πούμε, για παράδειγμα, να θεσμοθετηθεί δηλαδή αυτή η κατάσταση και να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν και το, η Γραμματεία του Συμβουλίου, καθώς και διεθνείς, περιφερειακές, ΜΚΟ και οι εμπειρογνώμονες, να είναι ένα φόρουμ ψηλού επίπεδου που θα πρέπει να φτάνει σε στόχους και στρατηγικές. Υπάρχει τέτοιο φόρουμ που προβλέπεται από την εξωτερική πολιτική της Ένωσης και θα ήταν μια μεγάλη προσθήκη στην αρχιτεκτονική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν θέλουμε δηλαδή να δούμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να έχουμε ένα συγκεκριμένο βήμα που θα ζητώνται λεπτομερώς κάθε χώρα χωριστά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ε, σας ρωτήσω. Θέλει κανείς το λόγο? γιατί αν δεν θέλει κανείς το λόγο, προτιμώ να περάσουμε αμέσως στο τρίτο μέρος της ακρόασής μας και να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στο δεύτερο μέρος για τις παρεμβάσεις τους, για την παρουσία τους εδώ, στις Βρυξέλλες και να παρακαλέσω τους προσκεκλημένους του τρίτου μέρους της δημόσιας ακρόασης να λάβουν θέση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Χάστινγκς να μας μιλήσει πρώτα εκείνος σε αυτό το πάνελ του τρίτου μέρους. Sorry, Okay, so Συνεχίζουμε λοιπόν συνάδελφοι. Θα δώσω πρώτο το λόγο στον κύριο Χάστινγκς που είναι θαμώνα σχεδόν στην Επιτροπή, πολύ συχνά τον προσκαλούμε. Είναι Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Θα Μα μιλήσει για το θέμα, χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων από άποψη προστασία τη ιδιωτική ζωή και προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ κύριε Κινγκαγκολ. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα για την πρόσκληση στη σημερινή δημόσια ακρόαση που έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε χρόνο να αξιολογήσουμε και να συζητήσουμε την εφαρμογή του χάρτη και να δούμε πώς ε, μπορεί ή θα έπρεπε να ε, πειράζει καλύτερα τους πολίτες ή να τους αγγίζει. Και χαίρομαι γιατί συμμετείχα σε αυτή τη συνεδρία. Σε δύο χρόνια μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον για τα θέματα των δικών μου αρμοδιοτήτων, του ιδιωτικού βίου και της προστασίας δεδομένων, ο δεσμευτικός νομικός χαρακτήρας ε, του χάρτη είχε νόημα και μεγάλη αξία. Πριν να ε, επεκταθώ στις εξηγήσει, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση το πώς ε, ε, η συμπερίληψη του χάρτη στη συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε τη νομική αρχιτεκτονική της προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη. Μία από τις καινοτομίες του χάρτη που πανηγυρικά ανακηρύχθηκε ως πολιτικό έγγραφο το Δεκέμβριο του 2000 ήταν η εισαγωγή ενός αυθυπόστατου δικαιώματος προστασίας δεδομένων στο άρθρο 8. Η διάταξη αυτή είχε στενή ε, συνάφεια με το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά ξεχωριστή εντολή. Έχουμε βασικές ε, ε, αρχές εδώ στις προστασίες των δεδομένων, δηλαδή τα δεδομένα θα πρέπει να τη χάνουν δίκαιες προστασίες και για συγκεκριμένους λόγους. Η επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται μετά από συνένεση του ενδιαφερόμενου ή με άλλη νομική βάση, βάση. Ο καθένα έχει δικαίωμα στην πρόσβαση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί για τον ίδιο και, το, και δικαίωμα διόρθωση αυτών. Και τέλο, η συμμόρφωση με του κανόνε αυτού θα υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή. Και μάλιστα, όπω δήλωσε σε πρόσφατη λομολογία ε, κατά της Γερμανίας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ύπαρξη ανεξάρτητης εποπτικής αρχής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο βασική συνιστόσα της προστασίας δεδομένων. Με την θέση ισχύ της Ηθικής Λισαβόνας, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων έχει ανακηρυχθεί σε βασική γενική αρχή τη κοινοτική νομοθεσία. Η συνθήκη τη Λισαβόνα όμω έκανε και κάτι παραπάνω. Το δικαίωμα σε προστασία δεδομένων είναι τα λίγα δικαιώματα του χάρτη που ε, συναντάται και τη συνθήκη για τη λειτουργία της, Ευρω... Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 16 θεσπίζει το δικαίωμα σε προστασία δεδομένων και δημιουργεί ξεχωριστή νομική βάση ε, της προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου έχουμε πλήρη προστασία, ε, πλήρη αρμοδιότητα, συγγνώμη, κοινοτική. Δεν χρειάζεται να επικαλέσουμε το άρθρο 51 αυτή η επανάληψη δίνει την σημασία που έχει, δείχνει τη σημασία που έχει η προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη της Λισαβόνα έδωσε μεγάλη όθηση για τη διαμόρφωση μια κουλτούρα προστασία δεδομένων και μια νοοτροπίας προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από το ίντερνετ και τι ε, ε, τεχνολογίε τη επικοινωνία και τη πληροφορία ε, καθιστούν σημαντικό αυτό το θέμα τη προστασία των δεδομένων γιατί τα δεδομένα πια βρίσκονται παντού και η επεξεργασία τους δεν γνωρίζει σύνορα. Ε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται την αναθεώρηση των ε, ε, κανόνων προστασίας δεδομένων προκειμένου να γίνουν πιο περιεκτικοί, πιο εύχρηστοι στην πράξη, πιο αποτελεσματικοί και λιγότερο περίπλοκοι προκειμένου να διασφαλιστεί και να αναβαθμιστεί το δικαίωμα υψηλής προστασίας των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτή την άποψη Πολλοί παράμετροι αναφέρονται στο άρθρο 8 του χάρτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα προστασία του πλαισίου προστασία δεδομένων για να εξασφαλίσει με καλύτερο τρόπο την αποτελεσματική λειτουργία των εποπτικών αρχών, των εθνικών και της κοινοτικής. Και φυσικά ε, να χαρακτηρίζονται αυτές οι υποπτικές αρχές από ανεξαρτησία. Ε, η, συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε άρδεν την αρχιτεκτονική προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε μια ε, και παρότρινε σε μια αναθεώρηση των ε, ισχυωσών κανόνων. Βέβαια, η έκβαση αυτής της αναθεώρησης θα χρειαστεί καιρό. Πάντως, με εφαρμογή του χάρτη τα τελευταία δύο χρόνια διαρωτόμαστε, είχε πραγματικά αποτελέσματα στην πράξη εφαρμογή. Νομίζω σίγουρα είχε τέτοια πρακτικά αποτελέσματα στην προστασία των δεδομένων. Θα σας αναφέρω δύο τέτοιε εξελίξεις στην τελευταία διετία. Καταρχήν, ε, νομολογία του ΔΕΚ στην ε, υπόθεση ΣΕΚΕ που αναφέρθηκε προηγουμένως στο Νοέμβριο του 2010. Και επίσης έχουμε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική ε, αποτελεσματικής εφαρμογής του χάρτη τον Οκτώβριο του 2010. Στην ε, ε, απόφαση την ομολογία ΣΕΚΕ, το δικαστήριο χρειάστηκε να απαντήσει το κατά πόσο ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαιτεί τη δημοσίευση των νόμων γεωργών που λαμβάνουν κονδύλια από το Γεωργικό Ταμείο συνάδει με το δικαίωμα στην ειδική σφαίρα και την προστασία των δεδομένων που κατοχυρώνει ο χάρτης. Είναι σημαντική αυτή η νομολογία και μάλιστα έχει και ευρύτερε συνέπειε γιατί ακυρώνει τη σχετική ε, κοινοτική διάταξη θεωρώντας την ασυμβίβαστη με το δικαίωμα ιδιωτικής σφαίρα και της προστασία των δεδομένων. Θεωρήθηκε ότι καταστρατηγούσε αυτή η διάταξη τα σχετικά δικαιώματα και μάλιστα το ΔΕΚ θεώρησε αυτό το, με, το μέτρο δυσανάλογο αυτή τη δημοσίευση δηλαδή. Μια και δεν ε, φάνηκε ότι ο νομοθέτης είχε προηγουμένως ε, διερευνήσει εναλλακτικά μέτρα, λιγότερο παρεμβατικά. Η νομολογία αυτή επιβεβαιώνει ότι ο νομοθέτης όταν πρόκειται να υιοθετήσει ένα δικαίωμα που επεμβαίνει στα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη θα πρέπει να κάνει μια μελέτη επιπτώσεων και προηγουμένως να διερευνήσει λιγότερο παρεμβατικά μέτρα και μέσω και να αιτιολογήσει την τελική επιλογή ο νομοθέτης λέω και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε δεν αποκλείεται μια τέτοια δημοσίευση των ονομάτων των γεωργών, αλλά επέμεινε το ΔΕΚ να είναι πολύ πιο προσεκτικό το θεσμικό όργανο για να εξασφαλίσει αναλογικότητα. Η νομολογία ΣΕΚΕ ε, ασθενίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και στηρίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην, στρατηγική της, στην ανακοίνωσή της για τη στρατηγική αποτελεσματικής εφαρμογής του χάρτη. Και αναφέρθηκε ότι ο χάρτης θα πρέπει να, αναφερθεί, να θεωρηθεί ως πηξίδα, όχι ως ε, ραδί, ως φόβητρο, αλλά ως πηξίδα. Επίσης, θα πρέπει να γίνει το τεστ της αναλογικότητας ε, ε, για την ε, θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων. Η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της τονίζει και την ανάγκη της εκτονιστέρων των υστέρων αξιολόγησης ε, υφιστάμενης νομοθεσίας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η εκτονιστέρων των αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας δεδομένων, γιατί εκεί ο νομοθέτης, ο Ευρωπαίος νομοθέτης, στην εποχή μετά του, την 11 Σεπτεμβρίου είναι παρεμβατικός. Έχουμε λοιπόν διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να γίνεται ε, το σύστημα αυτό ε, να περνάει από έλεγχο και από αξιολόγηση. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη τακτικής ε, παρακολούθησης και ενημέρωσης για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων. Με ένα μέτρο για, να, για ένα μέτρο που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια θα πρέπει να υποβάλλεται σε αξιολόγηση για να διαπιστώνετε κατά πόσο όντως είναι αποτελεσματικό και για το κατά πόσο συνιστά πραγματικά απαραίτητο και αποτελεσματικό μέτρο. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο του συνολικού αρχιτεκτονικού Και μάλιστα η αξιολόγηση και τη οδηγία για την κράτηση των δεδομένων, παρακράτηση δεδομένων θα πρέπει να αναφερθεί. Και η Κομισιόν το λαμβάνει αυτό σοβαρά υπόψη, γιατί ε, με βάση τι φιλοδοξίες της ανακοίνωση προσπαθεί να συγκεντρώσει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για να αποδείξει την, ανάγκη, την αναγκαιότητα για συγκεκριμένο νομοθετικό εργαλείο. Βέβαια στην πράξη είναι περίπλοκη αυτή η διαδικασία και αρκετά ε, χρονοβόρα γιατί δεν είναι και πολύ πρόθυμα τα κράτη-μέλη στη χορήγηση των στατιστικών στοιχείων που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως γίνεται αυτή η προσπάθεια και χαίρομαι που γίνεται, ελπίζω να επεκταθεί. Γιατί αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να βάλει τις προδιαγραφές για την αξιολόγηση και άλλων κοινοτικών εργαλείων που επηρεάζουν την ιδιωτική σφαίρα και την προστασία δεδομένων. Η νομολογία λοιπόν ΣΕΚΕ και η ανακοίνωση για το χάρτη δείχνουν ότι ο χάρτης τουλάχιστον στον τομέα προστασία δεδομένων και ιδιωτική ε, σφαίρα, είχε συγκεκριμένα αποτέλεσματα την τελευταία διετία και άμεσα για του πολίτε. Για παράδειγμα, δεν δημοσιεύονται πια τα ονόματα των γεωργών που λαμβάνουν ε, κοινοτικέ ε, επιδοτήσει. Και έμεσα έχουν αποτελέσματα για τους πολίτες μέσω των απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρεί ο νομοθέτης πριν υποβάλει ή θεσπίσει κάποια παρεμβατικά μέτρα. Επίσης, η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων που ξεκίνησε με το χάρτη θα έχει μεγάλο αντικτύπο στο μέλλον. Ως επόπτης, Ευρωπαίος επόπτης της προστασίας δεδομένων θα φροντίσω και θα μεριμνήσω στα πλαίσια των αρμοδοτήτων μου ε, ώστε τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και στο καθημερινό τους έργο αλλά και στις νομοθετικές προτάσεις να καθοδηγούνται από την πηξίδα του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και ευελπιστώ ότι θα συμβάλλω στην αποτελεσματική εφαρμογή του χάρτη και στα μελλοντικά χρόνια που περιλαμβάνουν σημαντικές προκλήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Χάστινγκς. Ε, ευχαριστούμε. Δίνομαι στο λόγο στον κύριο Πιέρ Μποσάν, διευθυντή της κοινωνικής πλατφόρμας. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, μια που είναι το τελευταίο πάνελ αυτό και δεν είναι πάντα εύκολο. Θα ήθελα να ανταλλάξω μαζί σας ε, απόψεις για το πώς μπορούμε να κάνουμε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη πιο αποτελεσματικό και θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα ε, σε αυτό το οποίο θεωρούμε τους αόρατους πολίτες του χάρτη. Πρώτα απ' όλα να σας παρουσιάσω την κοινωνική πλατφόρμα. Είμαστε ένα δίκτυο ευρωπαϊκών ΜΚΟ, 45 ΜΚΟ που εργάζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να αναφερθώ στις προϋποθέσεις πρόσβασης ε, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα παρουσιάσω εδώ πέρα άρα τέσσερα εμπόδια για να ασκήσει κανείς τα δικαιώματα του χαρτού του. Πρώτο είναι φτώχεια, δεύτερον απειρία, τρίτον διάκριση και τέταρτον παρεμπόδιση από τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή του χάρτη. Δεν είναι το θέμα μόνο να αναφέρουμε τα προβλήματα, θα ήθελα μαζί να ανταλλάξουμε απόψεις Το πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει το θεμελιώδη αυτό χάρτη και ειδικά τη σχέση μεταξύ των πολιτικών τη Ένωση και του χάρτη. Γιατί το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι να ε, κάνουμε μια διάκριση μεταξύ του χάρτη και των στόχων του χάρτη και του χάρτη ως μέσο, γιατί όλοι πιστεύουμε πως θέλουμε να εφαρμόσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει οπωσδήποτε μέσω του χάρτη ή μέσω μιας άλλης ευρωπαϊκής πολιτικής που θα στηρίξει το χάρτη. Θα ξεκινήσω με την ακραία φτώχεια. Δεν θέλω τώρα να κάνω μαθήματα γιατί όλοι εδώ μέσα ξέρουν ποιες είναι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Το 1998 είχαμε 18 εκατομμύρια φτωχούς και από ό,τι βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση τα πράγματα αυξάνονται. Πρώτον, είναι η πραγματικότητα. Δεύτερον, κάποια στιγμή και όταν ζούμε εδώ και στις Βρυξέλλες αλλά και έχουμε παραδείγματα από τα κρατη μπορούμε να βρεθούμε στην ιστορία. Θα αναφερθώ εδώ πέρα στην ΙΠΑ και στο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων που είπε το 1967 το εξής. Μετά από 13 χρόνια αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα. Είπε, αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα ξεκινούσα από τη φτώχεια. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή κάποιο είναι φτωχό, πάντα μιλάμε για την παγίδα της φτώχειας, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την παγίδα του νόμου. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Το ένα αφορά το Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή κάποιο είναι φτωχό και μπορεί να συμβεί στον καθένα όταν κάποιο χάνει το σπίτι του χάνει την ταυτότητά του, την κάρτα παραμονής. Μετά δεν μπορεί να ψηφίσει, δεν μπορεί να έχει κοινωνικά επιδόματα, χάνουν όλα τους τα δικαιώματα που αναφέρει ο χάρτης εδώ πέρα. Το δεύτερο παράδειγμα, και υπάρχει και στο site του Κοινοβουλίου, είναι ένα παράδειγμα, είναι κάτι που συνέβη στη Δανία. Το Δεκέμβριο του 2010 η αστυνομία πήγε σε ε, ένα άσυλο για αστέγους, μάζεψε όλους τους μη δανούς πολίτες και επειδή δεν μπορούσαν να συντηρηθούν στη Δανία, τους μάζεψε. Αυτό είναι παραβίαση του άρθρου 14 της συνθήκης που λέει μη διάκριση με βάση την εθνικότητα και βασίζεται μόνο στο κοινωνικό καθεστώς. Δηλαδή δεν ήταν επειδή ήταν αλλοδαποί και πολίτες της Ένωσης, αλλά επειδή δεν είχαν λεφτά και ήταν φτωχοί. Τι μας λέει αυτό, τι μας λένε αυτά δύο παραδείγματα, το Equinet λοιπόν το δίκτυο μας αυτό δείχνει πως ο κοινωνικός αποκλεισμός ε, οδηγεί σε μεγαλύτερη διάκριση και δεν μπορεί κανείς να ασκήσει τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Και έχει προτείνει η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τα ε, κοινωνικά δικαιώματα επίσης να μελετηθούν. Οπότε όταν είναι κάποιος στη φτώχεια δεν σκέφτεται καν την πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα. Οπότε τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 21 ε, που είναι διάκριση με βάση την κοινωνική διάσταση αλλά σκεφτείτε και το άρθρο 9 της συνθήκης που λέει πως ε, καθορίζοντας την πολιτική της η Ένωση θα λάβει υπόψη την ε, προώθηση της απασχόλησης, ε, την κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εκπαίδευση πρώτον. Δεύτερον, οι πολιτικές της Ένωσης, ε, η στρατηγική 2020. Τρεις από τους στόχους εκεί πέρα αφορούν την κοινωνική συμπερίληψη, τη φτώχεια, την εκπαίδευση και την απασχόληση. Αυτά λοιπόν τα πράγματα μπορούν να χρησιμοποιήσει Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν για να υποστηλήσουν στου ανθρώπου να βγουν από τη φτώχεια και να ασκήσουν τα θεμελιώδη του δικαιώματα. Αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα δεν είναι να παίζουμε με τα άρθρα του χάρτη, αλλά να δούμε ποιο είναι ο μηχανισμός που χρειάζεται έτσι ώστε οι άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια να έχουν θεμελιώδη δικαιώματα. Και ερχόμαστε έτσι εδώ πέρα στο δεύτερο φράγμα άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι η αναπηρία. Ανέφερα το άρθρο 26 που λέει πως θα πρέπει να υπάρχει ενσωμάτωση, αλλά εδώ και πολλά, για πολλά χρόνια μάλλον δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο και η Ένωση πρώτα απ' όλα. Μπορείτε να ζητήσετε από το Συμβούλιο να υιοθετήσει το άρθρο 19 της Οδηγίας για μη διάκριση στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Δεύτερον, μπορείτε να υποστηρίξετε την ε, πρωτοβουλία της Κομισιόν για τον νόμο περί αναπηρίας που θα προταθεί το επόμενο έτος. Αλλά εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που είναι η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόπων με αναπηρία. Γιατί, Γιατί η σύμβαση του ΟΗΕ που κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τι λέει. Δεν δίνει νέα δικαιώματα στους ανθρώπους με αναπηρία, προτείνει νομικούς μηχανισμούς για να μπορέσουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Και εδώ πέρα επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπα για τη φτώχεια, γιατί νομίζω πως το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο μπορούν να ξεκινήσουν να βρουν ένα νομικό μηχανισμό για το πώς οι φτωχοί θα μπορούν να έχουν θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε. Το τρίτο, ο τρίτος φραγμός θα ήθελα να αναφέρω είναι το άρθρο 21, οι διακρίσεις. Υπάρχουν διαφορετικά ζητήματα εδώ πέρα και για να επανέλθω στο παράδειγμα που ανέφερα στη ΣΥΠΑ, αυτό το οποίο έλεγαν πάντα ήταν πως τα δικαιώματα δεν αφορούν μόνο την νομοθεσία ή την εκπαίδευση. Είναι και τα δύο. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία μας, πρέπει να εργαστούμε μέσω της νομοθεσίας, αλλά να αλλάξουμε και την εκπαίδευση, το πώς εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους. Και αν δείτε την κατάσταση σε κάποια κράτη-μέλη, π.χ. στην Ιρλανδία, όταν οι ε, μαθητές που είναι γκέι και λεσβίες ε, υφίστανται ε, ε, παρενόχληση στα σχολεία, τότε πώς όταν θα μεγαλώσουν θα συμπεριφερθούν σύμφωνα με όσα λέει ο χάρτης. οπότε πρέπει να το δούμε αυτό από πλευρά διακρίσεων και εγώ θα ήθελα βεβαίως να σκεφτείτε κάτι εντός κοινοβουλίου και αφορά την υπηκότητα και βεβαίως αναφέρομαι σε υπηκόους τρίτων χωρών. Εάν Σκεφτείτε την αρχαία Ελλάδα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν πολίτες ήταν επίλυτες σε αυτή την πόλη. με τα κτλ. Έχουμε προχωρήσει πολύ. Σκεφτείτε τους σκλάβους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ανθρώπινα όντα. Αν σκεφτείτε τους μαύρους οι οποίοι μέχρι το 64 δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα οι γυναίκες ε, δεν είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν ε, τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε θα κάνουμε το βήμα έτσι ώστε οι άνθρωποι από τρίτες χώρες να μπορούν να έχουν θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως ε, πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο μέσος και όταν μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα να αφορούν τα ανθρώπινα όντα, όχι μόνο τους πολιτές της Ένωσης. Και το τέταρτο, το εμπόδιο, είναι η παρεμπόδιση από τα κράτη-μέλη και πρέπει να σκεφτούμε την ε, άμεση εφαρμογή της ε, χάρτας. Θα αναφέρω εδώ πέρα τη χώρα στην οποία μένουμε περισσότερο, που είναι το Βέλγιο, όταν μιλάμε για φτώχεια και πρόσβαση στα δικαιώματα. Το Κοινοβούλιο, Κομισιόν κτλ. Ε, έχουν δημοσιοποιήσει το χάρτη, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε είναι αποτελεσματικότητα στην άσκηση των δικαιωμάτων. Όταν λέει ένα κράτο μέλος ναι για να έχει κανείς κοινωνική ασφάλιση ε, θέλω να έχετε κατοικία ή άδεια παραμονής. Τότε το κοινοβούλιο βγάζει ένα ψήφισμα και λέει αυτό το οποίο κάνει το Βέλγιο είναι λάθος. Μπορεί να κάνει το εξή. Ότι χρειάζεσαι μετά το χ ή το ψ πράγμα για κοινωνική ασφάλιση. Πρέπει να σκεφτούμε νομικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να κατησχύει οποιασδήποτε εθνική νομοθεσία ε, χάρτη για να μπορούν οι άνθρωποι να ασκήσουν τα δικαιώματά του και να μην χρειάζεται να περιμένουν δεύτερο. Πάλι από το Βέλγιο. Ε, για το άσυλο. Δεν ξέρω αν ακούσα το βελγικό ραδιόφωνο σήμερα το πρωί, αλλά η υπηρεσία ασύλου τσακώνεται με την υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης. Τι λέει το Ομοσπονδιακό κράτος, λέει άστους εκεί πέρα και εγώ δεν έχω πόρους ανθρώπινους και δεν έχω πόρους ε, οικονομικούς. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στο Βέλγιο με δικαιώματα που τους δίνει ο χάρτης, θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτά άμεσα και θα πρέπει, δεν, είναι δυνατόν να τους κοροϊδεύουν από τον Άννα στον Καϊάφα. Τέλος, για τα σχόλια της Κομισιόν, για τις δύο υπηρεσίες, between EU policies and the Charter. And the, of was saying we should have clear separate... Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής εντολή μεταξύ της υπηρεσίας του Δουβλίνου και της Βιέννης. Ε, γιατί δεν συνεργάζονται. Γιατί να μην έχουμε μια κοινή έκθεση Βιέννη και Δουβλίνο για το πόσο ο μηχανισμός ε, της φτώχειας ε, να μπορέσει να παραμεριστεί για να ασκήσουν οι άνθρωποι τα θεμελιώδη του δικαιώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, Και τώρα θα δώσω το λόγο στην τελευταία μιλήτρια, την κυρία Τρέισι Γκόρτ, που είναι ανώτερο σύμβουλο πρωτοβουλία για τη δικαιοσύνη ε, του Ιδρύματο Ανοιχτή Κοινωνία. Σα ευχαριστώ. Ονομάζομαι Τρέισι Γκέρντ. Είμαι μέλος της πρωτοβουλίας ε, για την δικαιοσύνη του Ιδρύματος Ανοιχτή Κοινωνία. Καλωσορίζουμε την ευκαιρία μπορούμε να, να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας το έργο μας και να βρούμε καλύτερους τρόπους για να μπορέσουμε, μπορέσει να εφαρμοστεί ε, πιο ε, σωστά ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σήμερα θα σας μιλήσω λοιπόν για δύο ευρωπαϊκές περιπτώσεις ε, των οποίων έχουμε εστιάσει την προσοχή μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στην Τσεχική Δημοκρατία λοιπόν και μάλιστα μία υπόθεση έχουμε για τους Ρωμά και για την πρακτική που ακολουθούν να στέλνουν τα παιδιά των Ρωμά σε ειδικά σχολεία ε, λόγω της ε, προέλευσής τους. Και η περίπτωση αυτή μας δείχνει πόσο πολύ ε, παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ισότητας, της ε, ένταξης ε, και του σεβασμού. Τα βλέπουμε αυτά ως ενδεικτικά μιας ευρύτερης τάσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και συγχρειάζεται το Κοινοβούλιο να τα προσέξει αυτά. Καθώς βαθαίνει η κρίση του ευρώ και η ξενοφοβία αυξάνεται, οι Ρωμά σε ολόκληρη την Ήπειρο αισθάνονται στο πετσί τους την εχθρική κοινή γνώμη καθώς και τις ε, εχθρικές πολιτικές, κυβερνητικές πολιτικές. Ενθαρρύνουμε λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο να καταστήσει σαφή την αποφασιστικότητά του να, να, να καταπολεμήσει τις διακρίσεις κατά των φτωχότερων και των πιο ευάλωτων και να μην χρονοτριβεί. Ένας απλός τρόπος είναι ναι, εμένα, ο χάρτης υπάρχει ως νομική ε, υπέρμαχή του γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το, η νομοθεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο για κοινωνική αλλαγή και ως ένα μέσο για να στηριχτούν οι ιδέες από τον οποίων φτιάχτηκε η Ευρώπη παρόλο που οι ιδέες αυτές έχουν και αυτές τα όρια τους. Ωστόσο το μήνυμα είναι ότι ο χάρτης χρειάζεται να στηριχτεί με άλλους τρόπους, ιδιαίτερα πολιτική ενίσχυση και πίεση ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται σεβαστά και τηρούνται και εφαρμόζονται μάλλον στην πράξη. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να σας δείξω τρόπους ε, που αυτό είναι δυνατόν να γίνει χρησιμοποιώντας παραδείγματα. Καταρχήν να μιλήσω για την τσεχική δημοκρατία. Το 99 ο εκτελεστικός μας διευθυντή πήγε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 18 παιδιά στην τσεχική δημοκρατία. Τότε οι στατιστικές έδειχναν ότι τα παιδιά των Ρωμά ήταν, ε, ε, είχαν 27 φορές πιθανότητες περισσότερες από τα άλλα παιδιά να μπουν σε ειδικά σχολεία και τους, τους διδασκόταν ένα περιορισμένο, μια περιορισμένη ύλη. Από τη στιγμή που έμπαιναν σε ειδικά σχολεία ήταν σχεδόν αδύνατον να βγουν από αυτά και αυτή η παιδεία κάτω των προδιαγραφών περιόριζε τη ζωή τους και τις ευκαιρίες τους αργότερα. Οχτώ χρόνια αργότερα το 2007 κερδίσαμε την υπόθεση αυτή μάλιστα. Το, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε πως η Τσεχία παράνομα έκανε διακρίσεις κατά των ε, παιδιών των Ρωμά και, ενεργούσε ενάντια στα δικαιώματά τους στην ισότιμη παιδεία και διέταξε την Τσεχική Δημοκρατία να πληρώσει αποσημειώσεις σε όλα αυτά τα παιδιά καθώς και να θεσπίσει μέτρα ώστε να πάψουν οι διακρίσεις που βασίζονται στην εθνικότητα, στην εθνότητα καθώς και να διορθώσει όποια βλάβη είχαν υποστεί τα παιδιά αυτά στην Τσεχική Δημοκρατία. Βέβαια, Πεόρο απέχει η τσεχική δημοκρατία από την πλήρωση αυτή της νομικής υποχρέωσης και η ιδέα της παιδείας ε, είναι ε, παραμύθι για τα περισσότερα παιδιά Ρωμά στην τσεχική δημοκρατία. Και ενώ η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες, τουλάχιστον επί χάρτου, για να εφαρμόζει τις αποφάσεις αυτές, δεν βλέπουμε καμία κίνηση επιτόπου. Ενώ δηλαδή αναπτύσσει ένα πρόγραμμα δράσης για την ε, παιδεία, η εφαρμογή του στην ουσία είναι τελματωμένη. Το Υπουργείο Υποτίθεται ότι έχει λάβει μέτρα για να πάψει η διάκριση επί τη βάση εθνοτικής προέλευσης, αλλά είναι ανεπαρκή όλα αυτά. Η ισότητα δεν στηρίζεται συστημικά. Τα παιδιά Ρωμά δεν στηρίζονται για να πετύχουν στην κανονική εκπαίδευση και αυτό το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Επίσης, σχέδια για να δαπανηθούν ε, χρήματα της Ένωσης για την ισότιμη ε, ε, παιδεία και για την ένταξη των παιδιών αυτών στην βασική εκπαίδευση δεν έχουν εφαρμοστεί ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί. Ξέρουμε πως κάθε χρόνος που περνά χωρίς δράση ακόμα μια γενιά παιδιών μπαίνουν σε ένα αδιέξοδο μέλλον. Άρα λοιπόν ήρθαμε σε επαφή με την Επιτροπή των Υπουργών που επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους ενημερώσαμε ότι δεν έχει γίνει πρόοδος επιτόπου. Το ίδιο κάναμε και με τα αρμόδια σώματα του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και για την Επιτροπή για την εξάλληψη των διακρίσεων στην παιδεία και οι δύο ζήτησαν την ε, πάυση αυτού του συστήματος. Ελπίζουμε ότι θα ασκηθεί κατάλληλη πολιτική πίεση και θα γίνουν οι αλλαγές αυτές. Τώρα για την Ιταλία και για το θέμα όπου γνωρίζουμε πως η Επιτροπή σας ημερίζεται την ίδια θέση με μας, όπου οι κατασκηνώσεις Ρωμά απειλούνται με άμεση, άμεσο κλείσιμο και η Ρωμά με έξωση, ε, εδώ έχουμε έρθει σε επαφή με τους ε, νομάρχες Ρώμης, Νάπολης και Μιλάνου, οι οποίοι έλαβαν ε, την εξουσιοδότηση να ενεργήσουν με εξαιρετικά μέτρα, έκτακτα μέτρα, εκεί όπου υπήρχαν κατασκηνώσεις Ρωμά. Να κάνουν υπογραφή με συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων που ζούσαν σε αυτές τις κατασκηνώσεις ήταν Και επίσης έπρεπε να καταργηθούν αυτές οι κατασκηνώσεις και να δημιουργηθούν νέες. Βασικά η Ιταλική κυβέρνηση έτσι έφτιαξε μια βάση δεδομένων που μόνο για τους Ρωμά έτσι ώστε να μπορέσει να διαλύσει τις κατασκηνώσεις αυτές και να απελάσει τους Ρωμά. Παρά συγκεκριμένα αιτήματα οι νομάρχες δεν έδωσαν ποτέ τις κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες που χρησιμοποίησαν κατά το Ρωμά, ποια ήταν τα συστήματα που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της επιγραφής, ούτε έδωσαν πληροφορίες για το στον οποίο οι στόχοι της απογραφής αυτή επετεύθησαν. Και επίσης τα αιτήματα για διαγραφή όλων αυτών των στοιχείων ε, απορρίφθηκαν. Παρά τις ανησυχίες που εξέφρασε αυτή η Επιτροπή, η κατάσταση αυτή, η επίγουσα κατάσταση συνεχίζει να επικρατεί τρία χρόνια μετά. Και στην έκθεση του 2011 ο Επίτροπος Σάμεμπεργκ ε, πρότεινε να αλλάξει η εστίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί δηλαδή να έχουμε στόχο την ε, ε, απέλαση να έχουμε το στόχο την κοινωνική ένταξη όλων αυτών των ανθρώπων. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο εμείς και άλλες ε, ΜΚΟ εταίροι μας προσπαθήσαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει η δικασία επιπαραβίαση κατά της Ιταλίας για την παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ισχυριζόμαστε ότι τα μέτρα αυτά παραβιάζουν τρεις τομείς, προστασία δηλαδή δεδομένων, ισότητα ε, λόγω φύλου και η οδηγία της ηθαγένειας παραβιάστηκαν από την Ιταλία. Και θα δοθούν και οι σχετικές, τα σχετικά σχετική φάκελη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα για την Τσεχία έχει παραβιαστεί το δικαίωμα στην παιδεία, το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εδώ νομίζω πως η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει το πολιτικό της κύρος ώστε ο χάρτης να γίνει πραγματικότητα. Και θέλουμε να, σκεφτείτε, να σας ζητήσουμε να σκεφτείτε τα εξή. Για την Τσεχία θα θέλαμε να ζητήσετε μια κοινοβουλευτική ερώτηση στην ε, τσεχική κυβέρνηση. Καταρχήν ενημέρωση για την εφαρμογή της περίπτωσης στη AIDS καθώς και για τις στατιστικές για τα παιδιά Ρωμά και μη Ρωμά στα ειδικά σχολεία και έπειτα το πώ δαπανώνται τα ευρωπαϊκά διευθυντικά ταμεία για το στόχο τη συμπεριληψη των παιδιών των Ρωμά στην βασική παιδεία και κατά πόσο δαπανώνται όντω τα χρήματα αυτά για αυτό το στόχο. Επίση, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κομισιόν να ρωτηθεί για το τι γίνεται με τη χρήση των διευθυντικών ταμείων για τη χρήση ειδικών δομών στην Τσεχική Δημοκρατία έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τηρούνται και πληρούνται οι απαιτήσει τη απόφαση του ΔΕΚ. Επίσης θέλαμε να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει η διαδικασία επί κατά της Ιταλίας. Να ζητήσουμε επίσης ε, την διαγραφή προσωπικών των στοιχείων μέσω, που συλλέχθηκαν μέσω της απογραφής καθώς και να αποτίσει τη δέσμευση των Ιταλικών αρχών για παροχή αυτόνομων καταλημάτων για τους χιλιάδες Ρωμά που εκδιώχθηκαν κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης επίγουσης κατάστασης. Θα πρέπει επίσης να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πιο στενά με την πλατφόρμα για τους Ρωμά για τους οποίους ε, οι υποσχέσεις της συνθήκης της Λισαβόνας είναι ακόμα ένα μακρινό όνειρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γκάρτ. Η κυρία Γκόμες τώρα έχει το λόγο. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Χάστινγκς. Άκουσα την ομιλία σας και αναφέρθηκατε στην ανάγκη ανεξάρτητης εθνικής επιπτικής αρχής ε, για την ε, προστασία των δεδομένων. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από την ομολογία ΣΕΚΕ, για την απόφαση ΣΕΚΕ. Στην περίπτωση της χώρας μου, ε, έχει υπογράψει η κυβέρνηση της Πορτογαλίας διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ για το PNR, για τη μεταβίβαση δεδομένων προεξοφλώντας, προδικάζοντας αυτή που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν έγινε καν διαβούλευση με την Εθνική Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Και μάλιστα πριν την επίσημη έγκραση από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο έγινε σχετική δήλωση Μία δήλωση άλλωστε που αποτελεί κατάφορη παραβίαση και όχι μόνο του χάρτη θεμελιώδων δικαιωμάτων, αλλά και του ίδιου του συντάγματος της Πορτογαλίας. Υπάρχει λοιπόν Εθνική Εποπτική Αρχή και η δήλωση της ε, Εποπτικής Αρχής ήταν ε, κατηγορηματικότατη ως προς την ασυμβατότητα της συμφωνίας, διμερούς συμφωνίας και τον αντισυνταγματικό της χαρακτήρα. Ο Κάρλος Κόλιο, ο Ρούτα Βάρης και οι υποφαινομένοι κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου κατά της ε, συμφωνίας αυτής, που παρόλα αυτά όμως υπογράφηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εσείς έχετε δικαίωμα να κάνετε κάτι, να δράσετε, να αναλάβετε κάποια δράση κατά της πορτογαλικής κυβέρνησης. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δράσει. Και αναφέρω την περίπτωση αυτή της Πορτογαλίας, αλλά μπορεί να μην είναι η μοναδική ε, τέτοια περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο Ευρωπαίος Επόπτης δεδομένων, ο κύριος Χάστινγκς. Αν αυτή είναι η μοναδική σας ερώτηση, πολύ φοβάμαι ότι η απάντησή μου θα σας απογοητεύσει. Το γραφείο μου... Ε, εξασφαλίζει συμμόρφωση σε περίπτωση που υπάρχει κατάφορη παραβίαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνήθως ε, ε, παρέχουμε συμβουλές για νέες πολιτικές και για συμφωνίες PNR με τρίτες χώρες. Και με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να σας πω ότι πολύ συχνά οι συμβουλές που δίνουμε και οι συστάσεις λαμβάνονται υπόψη και μάλιστα πολύ συχνά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστερνίζεται τις συστάσεις μας και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Το ίδιο και το Συμβούλιο. Δέχεται κάποιες ε, ε, συμβουλές από εμάς ιδιαίτερα για θέματα PNR, TFTP, όπου αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Και παρενέβημεν σε πολλές περιπτώσεις. Ε, ασκήσαμε και προσφυγή στο ΔΕΚ. Και, και το ΔΕΚ έλαβε υπόψη τις θέσεις μας και τις συστάσεις μας, βλέποντας την περίπτωση της απόφασης κατά της Γερμανίας για την ε, ανεξαρτησία της Επιτικής Αρχής. Αλλά αυτά που συμβαίνουν στα εθνικά κοινοβούλια ε, ξεφεύγουν από τις αρμοδιότητες μας. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ε, γύρει προσφυγή επί παραβάση κατά συγκεκριμένη χώρα. Αλλά αν πρόκειται για μια συμφωνία που ετοιμάστηκε στο Συμβούλιο και υπευλήθη ε, σε εθνικό στα εθνικά κοινοβούλια για έγκριση, κάτι που συνέβαινε πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας, εκεί υπάρχει πρόβλημα που ίσως το διορθώνει όμως η θέση σε εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας, αλλά εγώ δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Ε, Εμεί συνεργαζόμαστε με εθνικούς επόπτες προστασία δεδομένων και με τον Πορτογάλο επόπτη και ρόλος μου είναι να εξασφαλίσω μια συνέπεια, συνάφεια όπου είναι δυνατόν. Αν υπάρχει παραβίαση, μη συμμόρφωση, το σημειώνουμε, αλλά δεν μπορώ εγώ να σας εξηγήσω κάτι παραπάνω. Κλείνω το μικρόφωνο δυστυχώς της κυρίας Γκόμες. Είπα PNR αλλά μπερδεύτηκα λάθος. Αφορούσε μεταβίβαση δεδομένων η συμφωνία σε περίπτωση υπόνοιας διάπραξης εγκληματικής ενέργειας. Τότε ίσως μπορεί να έχει συναυθεί διμερή συμφωνία μεταξύ Πορτογαλίας και τρίτης χώρας, είπα προκειμένου. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε πολύ συχνά συνάπτουν διμερώς συμφωνίες με χώρες και καμία από αυτέ δεν ήταν ικανοποιητική για να το πούμε διπλωματικά. Ευχαριστώ κύριε Χάστινγκ και επανέρχομαι στην εισηγήτριά μα τώρα, στην κυρία Πλασίκοβα Μπένοβα για να ανακεφαλαιώσουμε και να ολοκληρώσουμε τη δημόσια κρόση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Κίνγκα και θα αντλήσω τα συμπεράσματα από την δημόσια αυτή ακρόαση, μιλώντας όμως σλοβακικά, τη μητρική μου γλώσσα. Περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας και ευχαριστώ και για την κατανόηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους προσκεκλημένους που συμμετείχαν στα τρία πάνελ, στα τρία μέρη της δημόσιας ακρόασης, Ε, ε έλαβα, πήρε το δό σημειώσεις, συμπλήρωσα δέκα σελίδες στο τετράδιό μου με σημειώσεις από τη δημόσια ακρόση και θα ήθελα να επικεντρωθώ στα τέσσερα κυρίως θέματα που αναφέρθηκαν σχεδόν από όλους ε, τους ομιλητές, από όλους τους εμπειρογνώμονες. Καταρχήν να ξεκινήσω από κάτι που ανέφερε στο πρώτο μέρος της ε, δημόσιας ακρόασης η Άννα Γκόμες. Είπε ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και με τους εαυτούς μας και με... να δούμε πρώτα τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, ε, να συμμαζέψουμε τα του οίκου μας και μετά να ενδιαφερθούμε για το τι συμβαίνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές ήταν οι ενδιαφέρουσες ιδέες και πολλές οι προτάσεις που διατυπώθηκαν και θα προσπαθήσουμε τις περισσότερες να τις εφαρμόσουμε. Να αναφερθώ σε κάτι που επισήμανε κάποιος ομιλητής στο τρίτο μέρος, το θέμα των Ρωμά, της ε, μειονότητας των Ρωμά. Εγώ κατάγομαι από τη Σλοβακία, μια χώρα με πολυπληθή κοινότητα Ρωμά και έχουμε επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά. Uh, Τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τη μειονότητα των Ρωμά αλλά και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τώρα να πω και κάτι θετικό. Ε, σε, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το τελευταίο εξάμεινο το πιο συχνό ερώτημα που θέτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά τους Ρωμά. Mm. Αυτό είναι πολύ θετικό γιατί δείχνει ότι χρησιμοποιούμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να παροτρύνουμε την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη το ζήτημα των Ρωμά και να κάνει επιτέλους κάτι, να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Και όχι μόνο να λάβει τις αποφάσεις που θα μείνουν κενό γράμμα, αλλά να τις, να τις εφαρμόσει και εμπράκτος. για να υπάρξουν απτά αποτελέσματα και να επιληθεί το ζήτημα των Ρωμά. Οι χώρες που έχουν μειονότητα Ρωμά αντιμετωπίζουν ε, παρόμοια προβλήματα. Και το ίδιο ισχύει και για τις χώρες Κεντρικής Ευρώπης, τα πιο νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ε, χώρες που ήταν από τις ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε και υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα ένας εκπρόσωπος ε, της Επιτροπής. Περιμένουμε το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κρίμα που έφυγε στο μεταξύ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως ε, διαπιστώνουμε σοβαρές αδυναμίες στη συνεργασία με τις εθνικές αρχές όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και με τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και πολλά θετικά παραδείγματα αγαστής συνεργασίας και αυτά τα παραδείγματα θα πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε για να βρουν μιμητές και να αξιοποιούμε καλύτερα και τα κοινοτικά κονδύλια ώστε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα των Ρωμά. Δυστυχώ ε, υποχρεωνόμαστε και επαναλαμβάνουμε το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι να κάνουμε με, τη, τους Ρωμά και με τα προβλήματα του, των Ρωμά. Η... Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια υιοθετεί πρόγραμμα εργασίας, αλλά η κατάσταση αντί να βελτιώνεται επιδεινώνεται. Η λύση του προβλήματος στο Ρωμά θα πρέπει να δοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι μόνο εθνικό ζήτημα ή περιφερειακό. Υπάρχει και το ζήτημα της φτώχειας, της ένδυας του πληθυσμού Ρωμά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεριζώσουμε αυτή την εξαθλίωση γιατί η εξαθλίωση αντιμετωπίζει η κοινότητα του Ρώμα, ιδιαίτερα στις ε, νέες χώρες μέλη, στι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που έχουν σημαντική μειονότητα. Αν καταφέρουμε λοιπόν στην έκθεσή μας και περιλάβουμε και κάποιες προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εξαθλίωση, της μεγάλη φτώχεια των Ρωμά, τότε σίγουρα θα επηρεάσουμε θετικά την, το γενικότερο ζήτημα των Ρώμα. Εν συντομία τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο άλλα σημεία. Σίγουρα και εσείς παρακολουθείτε το έργο της Επιτροπής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα γνωρίζετε ότι ε, εξετάζουμε δύο πολύ επίμαχα θέματα το θέμα του PNR, των συμφωνιών PNR και το θέμα της, ε, του εντοπισμού Τη χρηματοδότηση από παράνομες ενέργειες, κυρίω από του, της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Είχαμε θέμα PNR με την Αυστραλία και τώρα τελευταία με τι Ηνωμένε Πολιτείε, Είναι επίμαχο, επαναλαμβάνω το θέμα, γιατί αφορά πολλές πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών. Και στη συζητήση στην Ολομέλεια είπαμε επανειλημμένως ότι στόχος μας είναι να προσπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και να προστατεύσουμε και τα προσωπικά δεδομένα των συμπολιτών μας. Από αυτή την άποψη, οι με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά είναι περίπλοκες και πολυσύθετες και επιμαχής, γιατί η έννοια της πράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι διαφορετική στις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μερικές φορές φαίνεται να υπάρχει δίλημα μεταξύ της ε, προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της δημοκρατίας. Υπάρχει μια αντιπαλότητα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί τα δύο θέματα να τα συνδυάσει. Και ναι με να καταπολεμήσει την τρομοκρατία, χωρίς όμως να θυσιάσει σε αυτόν τον αγώνα την προστασία των δεδομένων. Θα είναι πάντως ισχυρή συζήτηση για την επίμαχο το θέμα. Και ένα τελευταίο σημείο τώρα, όπως ξέρετε... Εδώ εξετάζουμε όχι μόνο το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά οργανώσαμε αυτή την ακρόαση για να προετοιμαστούμε καλύτερα στην εκπόνηση της ετήσιας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. όλη αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα επηρεάσει και το περιεχόμενο αυτής της ε, ετήσιας έκθεσης που θα καταρτήσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλήξει στη μορφή που θα δώσουμε στην έκθεση, αλλά είμαι βέβαιη ότι οι συνάδελφοι θα δείξουν συνεργάσιμο πνεύμα προκειμένου να υιοθετήσουμε μια λύση που θα είναι αξιόπιστη όχι μόνο για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά κυρίως ε, θα ικανοποιήσει τους συμπολίτες μας. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να δουν στην αιτήσια αυτή έκθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μια απόδειξη ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι αξιόπιστη, μπορούν να υπολογίζουν σε αυτή γιατί είναι μια επιτροπή που προασπίζει τα δικαιώματά τους. Πάντως εγώ θα σπεύσω να εκπονήσω την έκθεσή μου και θα σας τη μοιράσω περιμένοντας τις αντιδράσεις σας και τις δικές σας προτάσεις. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω από σας που είστε εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχετε κι εσείς και να μας βοηθήσετε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να μην αναζητήσουμε τα σημεία διχόνοιας και διχασμού, αλλά τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή και τη συμβαστική λύση. Ευχαριστούμε Μόνικα, αναμένουμε την έκθεσή σου και αναμένουμε να συνεργαστούμε και όλα. Σε ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Σε ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και όσους μας άκουσαν. Ευχαριστώ τη γραμματεία και τους διερμηνείς. Κλείεται η συνεδρίαση. Ε, καλό σας βράδυ.